Dear colleagues, please be seated so that we can... Καθίστε αγαπητοί συνάδελφοι για να ξεκινήσουμε. Για να προλάβουμε να θέσουμε και ερωτήσεις όπως όλοι επιθυμείτε. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε με το σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης ε, που είναι οικονομικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Μίκα Λίντιλα, πρόεδρο του ΕΚΟΦΗΝ και Υπουργό Οικονομίας της Φινλανδίας. Σας καλωσορίζουμε κύριε Υπουργέ. Όπως όλοι γνωρίζετε, ο κ. Λίτιλα ανέλαβε ε, την ε, Προεδρία του Συμβουλίου Κοφίν την 1η Ιουλίου και χαιρόμαστε που δεχτήκατε την πρόσκλησή, σας, την πρόσκλησή μας να παρουσιάσετε τις προτεραιότητες της Φινλανδικής Προεδρίας. Η δράση για την κλιματική αλλαγή είναι μία από τις προτεραιότητες της Φινλανδικής Προεδρίας και η βιώσιμη ανάπτυξη και οι πρωτοβουλίες για τη διευκόλυνση της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος είναι στο προσκήνιο των προτεραιοτήτων σας. Είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν και ερωτήσεις και για άλλους τομείς βέβαια. Όπως γνωρίζουμε η Φινλανδική Προεδρία λαμβάνει χώρα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο λόγω των ευρωπαϊκών εκλογών και του διορισμού της νέας επιτροπής. Προσβλέπουμε σε καλή συνεργασία με τη Φινλανδική Προεδρία για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ω συνήθω, η σημερινή ανταλλαγή απόψεων περιλαμβάνει και έναν οικονομικό διάλογο με, μέσα στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση, στο γενικότερο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Υπενθυμίζω τι γενικέ αρχέ για την ανταλλαγή απόψεων. Θα δώσω το λόγο σε εσά καταρχήν κύριε Υπουργέ για 10 λεπτά να κάνετε μια εισαγωγική παρέμβαση και μετά θα έχουμε κύκλους ερωτήσεων και απαντήσεων. Ερωτήσεις και απαντήσεις ε, πέντε λεπτών ε, για όλες τις ε, κοινοβουλευτικές ομάδες και ενδεχομένως με δευτερολογία αν το επιτρέπει ο χρόνος και μετά θα ακολουθήσουν και άλλοι γύροι ερωτήσεων. Σας δίνω το λόγο για μια πρώτη εισαγωγική παρέμβαση περίπου 10 λεπτών όπως είπαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, ε, είναι τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω εν συντομία τις οικονομικές, χρηματοπιστωτικές ε, και δημοσιονομικές προτεραιότητες της Φινλανδικής Προεδρίας. Στη συνέχεια θα είμαι στη διάθεσή σας για τις ερωτήσεις σας. Βρισκόμαστε σε κρίσιμη εποχή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει υιοθετήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για τα επόμενα πέντε χρόνια. Στοχεύουμε σε μία όσο το δυνατόν ομαλότερη μετάβαση στον επόμενο θεσμικό κύκλο και θα συνεργαστούμε στενά με τη Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι εργασίες μας στον τομέα του ΕΚΟΦΗΝ εμπίπτουν στις τρεις βασικές προτεραιότητες της Προεδρίας μας. Καταρχήν, θα προωθήσουμε την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, στοχεύουμε σε φιλόδοξη πρόοδο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Και τρίτον, θα επιδιώξουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες της Ευρώπης εναντίον των εσωτερικών και εξωτερικών απειλών. Προωθώντας αυτές τις δραστηριότητες ως προτεραιότητες, θα επιδιώξουμε να ενισχύσουμε την τήρηση των κοινών αξιών μας και του κράτους δικαίου. Ξεκινώ με την πρώτη προτεραιότητα, ανταγωνιστικότητα και συνοχή. Μια ανταγωνιστική Ευρώπη εξαρτάται από εσωτερικές αγορές που λειτουργούν σωστά, με κεφαλαιαγορές που έχουν βάθος, μια ολοκληρωμένη τραπεζική ένωση και ένα ισχυρό πλαίσιο επίλυσης κρίσεων. Όσον αφορά την Ένωση κεφαλαιαγορών, θα συνεχίσουμε τις εργασίες για τα θέματα που εκκρεμούν, συμπεριλαμβανομένης ε, της ανάκαμψης και εξυγίανσης κεντρικού συμβαλωμένου και των προτάσεων για τη συμμετοχική χρηματοδότηση. Παράλληλα, θα ξεκινήσουμε εργασίες προς ένα νέο οδικό χάρτη για την επόμενη φάση της Ένωσης κεφαλαιαγορών. Όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση, έχουμε δεσμευθεί ότι θα καταβάλουμε προσπάθειες για τεχνικές εργασίες για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων. Προγραμματίζουμε επίσης να συνεχίσουμε τις εργασίες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η πρόταση σχετικά με τις δευτερεύουσες αγορές για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι έτοιμη για τους τριμερείς διαλόγους και χρειάζεται και περαιτέρω εργασία στο Συμβούλιο για την ανάκτηση των πρόσθετων ασφαλιών και εγγύησεων. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματικά. Αυτό συμπεριλαμβάνει εργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος υποστήριξης μεταρρυθμίσεων και στο χρηματοδοτικό και δημοσιονομικό μέσο της Ευρωζώνης, όπου θα συνεργαστούμε στενά με το Eurogroup. Συνεχίζονται οι εργασίες και για διάφορα άλλα νομοθετικά κείμενα για να ολοκληρώσουμε την αναθεώρηση της συνθήκης του ESM. Στο πλαίσιο ε, της αναθεώρησης της οικονομικής διακυβέρνησης, προγραμματίζουμε να γίνει μια συζήτηση για τη λειτουργία του δημοσιονομικού μας πλαισίου. Αυτό θα αποτελέσει σημαντικό θέμα στην άτυπη συνάντηση ΕΚΟΦΗΝ την επόμενη εβδομάδα. Και από αυτή τη συζήτηση μπορούν να προκύψουν σχόλια που θα χρησιμοποιήσει η Επιτροπή στην αναθεώρηση του πλαισίου. Ένα δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα φορολογίας είναι κέρια σημασίας για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή. Θα προωθήσουμε την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών. Η καταπολέμηση αυτή διεξάγεται σε παγκόσμιο επίπεδο και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συνεργαστούν στενά με τις χώρες του ΟΣΑ για την αναζήτηση συνολικών λύσεων. Ένα απλό και αποτελεσματικό σύστημα ΦΠΑ που να μπορεί να μείνεται κατά της απάτης είναι ουσιαστικό για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και για την προστασία των φορολογικών εσόδων. Θα προωθήσουμε λοιπόν τις συζητήσεις για τη δέσμη μέτρων για το οριστικό καθεστώς ΦΠΑ και σκοπεύουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία και για τις υπόλοιπες προτάσεις που βρίσκονται επιτάπητος για το ΦΠΑ. Θα συνεχίσει επίσης και η σχετική δουλειά στο πεδίο των ειδικών φόρων κατανάλωσης. Θα συνεχίσουμε τις τεχνικές συζητήσεις για την κοινή βάση φορολογίας εταιριών όσον αφορά την παγκόσμια εισφορά επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, όταν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών που συμμετέχουν, θα προωθήσουμε τις σχετικές εργασίες στο Συμβούλιο. Η επόμενη προτεραιότητά μας είναι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα βασίζεται σε οικονομικά κίνητρα και δημοσιονομικούς πόρους. Θα επιδιώξουμε μια ευρεία συζήτηση για το πώς μπορούν να ενσωματωθούν καλύτερα τα θέματα που έχουν σχέση με το κλίμα στο έργο του ΕΚΟΦΗΝ και θα χρησιμοποιήσουμε την εργαλειοθήκη που έχουμε στη διάθεσή μας για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Θέλουμε να αναπτύξουμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα σχέδιο εργασίας για τους Υπουργούς Οικονομικών σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Θα χρησιμοποιήσουμε για αυτό το σχέδιο εργασιών ε, το έργο που έχουν κάνει οι Υπουργοί Οικονομικών στο πλαίσιο του Συνασπισμού Υπουργών Οικονομικών για την Κλιματική Δράση που δημιουργήθηκε τον Απρίλιο ε, και του οποίου είμαι συμπρόεδρος μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών της Χιλής. Οι συνεχιζόμενες εργασίες ε, για το βιώσιμο πλαίσιο χρηματοδότησης και την ταξινομία του είναι επίσης πολύ σημαντικές και θέλουμε να τις προωθήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Τέλος, θα δρομολογήσουμε και μία συζήτηση για την φορολόγηση της ενέργειας στην Ευρώπη ως τμήμα της προσπάθειας προς μια Ευρώπη με ουδέτερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Και αυτό με φέρνει στην τρίτη και τελευταία προτεραιότητα στον τομέα του ΕΚΟΦΗΝ, που είναι η ασφάλεια. Το περιβάλλον μας ως προς την ασφάλεια αλλάζει συνεχώς. Προκύπτουν απειλές σε μορφές που είναι πιο δύσκολο να εντοπίζονται. Υπάρχει παραπληροφόρηση, υπάρχουν κυβερνοαπειλές και άλλες μορφές. Τέτοιου είδους υβριδικές απειλές είναι φθηνές ως προς το κόστος, έχουν χαμηλό κατόφλι χρήσης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να στοχεύσουν κάποια ευάλωτα σημεία μας, να δημιουργήσουν αμφισημεία ή να εμποδίσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων θα αρχίσουμε συζητήσεις για την αντοχή των χρηματοπιστωτικών υποδομών μας έναντι των υβριδικών απειλών και αυτό θα το ξεκινήσουμε στην άτυπη συνάντηση ΕΚΟΦΗΝ την επόμενη εβδομάδα. Σκοπεύουμε να επιδιώξουμε τη συνειδητοποίηση του θέματος αυτού την ευαισθητοποίηση όλων και να εντοπίσουμε πιθανούς τομείς περαιτέρω ενεργειών. Στον τομέα της ασφάλειας, η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας θα είναι ένα από τα βασικά θέματα της Προεδρίας μας. Θα ζητήσουμε από τους Υπουργούς να συζητήσουν το θέμα αυτό με βάση τις σχετικές εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε να υιοθετηθούν συμπεράσματα συγγνώμη, από το Συμβούλιο για ένα στρατηγικό θεματολόγιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τέλον, τέλος, ε, κέρια σημασία για την ασφάλεια είναι το θέμα της πρόληψης της ε, ανεξέλεγκτης μετανάστευσης. Οι εργασίες της Ευρωπαϊκής ε, Χρηματοπιστωτικής Αρχιτεκτονικής για την Ανάπτυξη είναι σημαντικό τμήμα για την αντιμετώπιση των ριζικών αιτίων της μετανάστευσης. Αυτό θα δρομολογηθεί τον Οκτώβριο με βάση τις συστάσεις της ομάδας των σοφών. Αυτά είχα να σας πω και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Μόνο 30 δευτερόλεπτα ξεπεράσατε το χρόνο σας. Αυτό είναι ρεκόρ για εδώ. Για να δούμε Μήπως οι Γερμανοί μπορούν να σπάσουν αυτό το ρεκόρ καλύτερα. Εγώ θα πάρω το λόγο τώρα. δικό μου είναι το πρώτο σλότ. Δεν έχω μιλήσει πολύ σήμερα. Σίγουρα θα συζητήσουμε πολύ για την κλιματική αλλαγή. Θα υπάρξουν πολλές ερωτήσεις. Γι' αυτό εγώ θα επικεντρωθώ σε διαφορά άλλα ζητήματα. Φορολόγηση. Χαίρομαι που άκουσα ότι αποτελεί προτεραιότητα για σας. Θα ήθελα όμως να καταλάβω σε περισσότερες λεπτομέρειες πόσο μακριά μπορείτε να πάτε. Φαντάζομαι ότι όλα τα θέματα φορολόγησης ε, δεν έχουν την ίδια φύση, αλλά είναι νευροζώνη αλλά όχι. Θα μπορούσατε να μας πείτε περισσότερα για την μεταρρύθμιση από την οποία θα εποφεληθεί πολύ η οικονομία. Πώς θα ξεμπλοκάρετε τη σημερινή κατάσταση, γιατί δεν γίνεται πρόοδος, δεν υπάρχει πρόοδος. Το δεύτερον, για το CCCTB, για τη φορολογική βάση. Από ό,τι καταλαβαίνω θέλετε να συνεχιστεί η τεχνική συζήτηση. Δεν ξέρω πόσο μακριά μπορεί να πάει. Οπότε θέλω να μου πείτε σε τι βαθμό πιστεύετε ότι υπάρχει περιθώριο να προχωρήσει η ενισχυμένη συνεργασία σε αυτό το τομέα. Και το τελευταίο, η ψηφιακή φορολόγηση. Πριν από μερικούς μήνες έκλεισε ο φάκελος γιατί το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να πετύχει συμφωνία. Οπότε να ρωτιέμαι, μήπως θα έπρεπε να ξανανοίξει η συζήτηση γι' αυτό και να το ξαναδούμε το θέμα. Γιατί η συμφωνία αυτή δεν προσθέτει τίποτα τελικά. Οπότε αυτά είναι τα θέματα που θέλω να ξέρω. Kiitoksia. Sorry, I... Στα φιλανδικά θα απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ για τις ε, ερωτήσεις σας, Πρόεδρε. Το πρώτο έχει να κάνει με το IT, ε που αποτελεί μία από την πρώτη ερώτηση για το ΦΠΑ. Και θέλω να ακούσω περισσότερα. Ξέρω ότι έγινε δουλειά πολύ από τη Ρουμανική Προεδρία καταρχήν για νομοθετική πρόταση και στόχος μας είναι να βελτιωθεί το τρέχον σύστημα ΦΠΑ. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ ιδιαίτερα εδώ στην πρόταση για τη συλλογή δεδομένων από τις υπηρεσίε πληρωμών. Όταν θα έχουμε αυτά τα δεδομένα θα μπορέσουμε να προετοιμαστούμε πολύ καλύτερα. Οι αρχές δηλαδή προκειμένου να εντοπίσουν τις απάτες που γίνονται στον τομέα του ΦΠΑ. Και έτσι θα βοηθηθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρόκειται για πρόταση η οποία έχει να κάνει με τις εξαιρέσεις, με τις παρεκκλήσεις για τα στρατιωτικά ζητήματα, για το στρατιωτικό εξοπλισμό δηλαδή. Ιδιαίτερα για τη φορολογική βάση και για το διασυνοριακό εμπόριο επίσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Υπάρχει και το θέμα της ψηφιακής ε, φορολόγησης. Είναι μια μεγάλη πρόκληση. Είναι στην ημερήσια διάταξη του G20 και η Φιλανδία που έχει την Προεδρία θα προσπαθήσει να επιταχύνει τη διαδικασία στο Συμβούλιο. Σημείο κίνησή μα είναι ότι οι χώρε μέλη πρέπει να βρουν μία λύση που να μπορούμε να την συμπεριλάβουμε στα εθνικά καθεστώτα. Να είναι κάτι το οποίο είναι συμβατό δηλαδή με τα όσα ισχύουν στις χώρες μέλη, χωρίς βέβαια να απειλείται η οικονομική ανταγωνιστικότητα. Παρακολουθούμε λοιπόν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις συζητήσεις και στον ΩΣΑ και μεταφέρουμε τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές έχουν. Όσον αφορά τώρα την κοινή βάση. Εδώ, τη φορολογική κοινή βάση, εδώ συνεχίζουμε το έργο σε τεχνικό επίπεδο βάσει των όσων έχουν κάνει οι προηγούμενες προεδρίες. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που απαιτούν βέβαια και πολιτική τοποθέτηση για να προχωρήσουμε. Δηλαδή σε τι βαθμό θα προχωρήσουμε, αν θα πρόκειται για όλους τους φορολογούμενους, αν προτείνουμε φορολογικά κίνητρα και πώς θα αντιμετωπίσουμε τις διατάξεις που ήδη υπάρχουν στην οδηγία για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τη σχέση με το έργο του ΟΣΑ. Ένα λούμα τώρα εκ μέρους ε, των σοσιαλιστών. Παρακαλώ. Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, πολύ χαίρομαι που σας βλέπουμε εδώ σήμερα. και συγχαρητήρια στο πρόγραμμα της Προεδρίας σας, το οποίο βρίσκω ότι είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο και είναι πολύ καλό γιατί περιλαμβάνει και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Και χαίρομαι που αναφέρεστε επίσης την καταπολέμηση της νομοποίησης ε, χρημάτων ε, από παράνομες δραστηριότητε. Η φορολόγηση είναι από τα δύσκολα ζητήματα το οποίο όμως θα πρέπει να εξετάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλω να έρθω στο θέμα των ψηφιακών επιχειρήσεων και την ψηφιακή φορολόγηση, γιατί αυτό είναι το μέλλον. Αυτό θα μας απασχολήσει και στο μέλλον και θα θέλαμε να δούμε συγκεκριμένα αποτελέσματα σύντομα. Διαπιστώσαμε ότι ο Γάλλος Πρόεδρος και ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο κ. Μακρόν και Τραμπ, συμφώνησαν για την φορολόγηση των ψηφιακών επιχειρήσεων. Έχετε εσείς πληροφορίες για την συμφωνία αυτή και είσαστε έτοιμος να κάνετε συγκεκριμένες προτάσεις για το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Επίσης, κάτι άλλο που διάβασα σε εφημερίδες σήμερα ότι είσαστε από τους τρεις πιο δημοφιλείς πολιτικούς στη χώρα σας. Ελπίζω να συνεχίσετε να είσαστε εξίσου δημοφιλείς και μετά από το εξάμεινο της Φιλανδικής Προεδρίας. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χανελούμα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο τελευταίος Υπουργός Οικονομικών είχε ήδη ασχοληθεί με αυτό το θέμα της Ρουμανίας. Όσον αφορά την ψηφιακή φορολόγηση, πρέπει να σας πω ότι δεν γνωρίζω καλά ε, το σύνολο των θεμάτων που συζήτησαν οι δύο πρόεδροι, αλλά για την ψηφιακή φορολόγηση σίγουρα η λύση είναι συνολική. Πρέπει να είναι συνολική για να είναι και αποτελεσματική οι λύσει στα φορολογικά ζητήματα πρέπει να εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Και κάτι που είναι ζωτική σημασία για μας είναι να ακολουθούμε, να παρακολουθούμε τι γίνεται στον ΩΣΑ, έτσι ώστε το Συμβούλιο από τη δικιά του την πλευρά να μπορεί γρήγορα να δράσει για να προτείνει λύση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο λειτουργεί βάσει συμφωνιών στις οποίες καταλήγει το σύνολο των χωρών μελών. Παίρνει χρόνο, όντως, καθυστερεί. Αλλά άμα δούμε τι γίνεται σε διεθνές επίπεδο, αν δούμε ποιος είναι ο ρυθμός εκεί, όπως το έχω πει και νωρίτερα, το βασικό είναι να παρακολουθούμε την προετοιμασία του έργου που γίνεται στον ΩΣΑ. Ευχαριστούμε. Ε, Ρουγκαριγκάνο, Ρινιού. Ευχαριστώ πολύ. Είναι χαρά για μας να, έχουμε ένα μέλος αδελφού κόμματος κοντά μας και σας συγχαίρω για τα καθήκοντά σας. Αναγνωρίζουμε τα καθήκοντα και τις προκλήσεις που τίθενται στην Προεδρία σας σε δύσκολη εποχή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μας έχουν επίσης εντυπωσιάσει οι προτεραιότητες που έχει θέσει η Προεδρία σας. Ένα πληρέστατο, μια πληρέστατη δέσμη μέτρων ε, που μας ικανοποιεί και χαιρόμαστε που το βλέπουμε. Ε, μία από τις μεγάλες προκλήσεις είναι η κατάσταση σε σχέση με το Brexit, όπως εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Ε, έχω καταρχήν μια πολύ απλή ερώτηση. Ποιες είναι οι διαπραγματεύσεις με, με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αυτή τη στιγμή. Πρόσφατα ελέγχθη ότι γίνονται σημαντικές πρόοδοι. Δεύτερον, ποια είναι η δική σας αξιολόγηση για το επίπεδο ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης για το ενδεχόμενο αυτού του σοκ εάν συμβεί το Brexit, ιδίω αν είναι ένα σκληρό Brexit χωρίς συμφωνία. Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την οικονομική σταθερότητα και την ανάπτυξη και ποια είναι τα μέτρα οικονομικής διακυβέρνησης και οικονομικών αποφάσεων, ποια είναι τα μέτρα που προτίθεστε να λάβετε και που νομίζετε ότι πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να είμαστε έτοιμοι εάν προκύψει ένα τέτοιο σκληρό Brexit που μπορεί να υπάρχει τώρα στον ορίζοντα με βάση τις απειλές του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Kiitoksia kysymyksestä. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Δυστυχώς, πρέπει να σας πω ότι το Brexit δεν είναι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ. Και βέβαια, εύχομαι να υπάρχει μια συμφωνία. Στον τομέα του ΕΚΟΦΗΝ, από όσο γνωρίζω, έχουμε εντοπίσει όλους τους δυνητικούς κινδύνους που συνδέονται με ένα τέτοιο ενδεχόμενο ξεκινώντας από την οικονομική ανάπτυξη και όπως σας είπα και πιο νωρίς, δεν είναι αρμοδιότητα του, του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ το Brexit. Επόμενος ομιλητής εκ μέρους των Πρασίνων, Βίλεν Ιμίστο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζουμε ότι θα καθοδηγήσετε και τη φινλανδική οικονομία με ε, συνετό τρόπο και έχω κάποιες ερωτήσεις για την κλιματική αλλαγή. Είναι ευρείες οι προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Φινλανδική Προεδρία έχει φιλόδοξους στόχους ε, για ε, την κλιματική αλλαγή μέχρι το 2025 και για τον τομέα της φορολογίας και της οικονομικής πολιτικής υπάρχει κάποια αντίφαση μεταξύ των δύο αυτών στόχων. Δηλαδή το επίπεδο φιλοδοξίας που έχετε ε, για τους κλιματικούς στόχους, για τη φορολογία και για την οικονομική πολιτική, πώς μπορείτε να τα συνδυάσετε. για τη χρησιμοποίηση της ταξινομίας για βιώσιμη, βιώσιμα οικονομικά, ε, ποια είναι ε, η γνώμη της Φιλανδικής Προεδρίας. για να μπορέσουμε να κινηθούμε προς ένα βιώσιμο μέλλον ε, και οικονομικά και περιβαλλοντικά. Και δύο συγκεκριμένα θέματα, οι επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα είναι το ένα, τα διεθνή σχέδια δράσης για το κλίμα και για δράσεις σχετικές με το κλίμα, ε, που τα κράτη-μέλη πρέπει να υποβάλουν σχέδια για τον περιορισμό των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα, αλλά πολύ λίγα έχουν γίνει. Θα κάνει κάτι η Εθνική Προεδρία για να περιοριστούν οι επιδοτήσεις ε, που είναι 55 δισεκατομμύρια ε, ευρώ το 2016, αρκετά υψηλό επίπεδο. Και κάτι άλλο, ο ΣΑ ζήτησε να αυξήσουμε τους πράσινους φόρους. Η Φινλανδία έχει κάνει αρκετά σε αυτό το επίπεδο, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ χαμηλή φορολογία για κάποια ενεργειακά προϊόντα. Τα επίπεδα φορολογίας ε, για συγκεκριμένε μορφέ ενέργεια είναι ένα θέμα που θα μπορούσε να εξετάσει η Προεδρία σα για να μπορέσουμε να έχουμε πράσινη φορολογία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί παραθυράκια στο σύστημα που θα μπορούσε να οδηγήσουν σε ένα λιγότερο αποτελεσματικό σύστημα πράσινη φορολόγηση. Ευχαριστώ. ilmastonmuutos ja sen vastainen toiminta on Suomen keskeinen prioriteetti. Για την κλιματική αλλαγή και για την βιώσιμη χρηματοδότηση, θέλω να πω ότι αυτή είναι ε, ε, συνδεόμενη ε, στόχη και ο σκοπός της βιώσιμης των βιώσιμων οικονομικών είναι να μπορέσουμε να έχουμε υποστήριξη προς μια πιο πράσινη και ουδέτερη ως προς τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος οικονομία. Αυτά αποτελούν προτεραιότητες για τη Φινλανδία και χαίρομαι διότι πολλοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί έχουν αρχίσει ε, να κατευθύνονται προς τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά. Μια τάση που υποστηρίζουμε. Όσον αφορά την ταξινομία, Ελπίζω ότι θα έχουμε ένα κοινό πρότυπο για να μπορέσουμε να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο το συντομότερο δυνατόν. Η ταξινομία θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη σωστά και χρειαζόμαστε μια καλή πρόταση. Είναι πιο σημαντικό το να έχουμε μια καλή πρόταση. Η ποιότητα λοιπόν έχει εδώ σημασία. Και αυτό θα εξυπηρετήσει τους στόχους μας σχετικά με οικονομία ουδέτερη ως προς τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Τώρα, όσον αφορά τη φορολογία, και αυτό είναι σημαντικό θέμα όταν μιλάμε για την κλιματική αλλαγή και την καταπολέμησή της. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις δράσεις μας και σε εθνικό επίπεδο, παρότι δεν εκπροσωπώ ε, τη Φινλανδία αυτή τη στιγμή, αλλά την Φινλανδική Προεδρία. Έχουμε, μπορώ να σας πω ότι έχουμε εφαρμόσει στη Φινλανδία σε εθνικό επίπεδο ε, κάποια μοντέλα για την ε, φορολογία και είναι θέματα που θα είναι στο άτυπο συμβούλιο, στην ημερήσια διάταξη του άτυπου συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ. Ο κύριος Γκούνερ Μπέκ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω θερμά στη σημερινή μας συνεδρίαση. Θα ήθελα να αναφερθώ λιγάκι στο θέμα της ψηφιακή φορολόγηση. Η δική μας η πολιτική ομάδα, η ID, στηρίζει σε μεγάλο βαθμό την αρνητική στάση της Φινλανδικής Προεδρίας για το θέμα αυτό. Όμως στην έκθεση που έχετε συντάξει, τη γραπτή, εκεί αναφέρεστε στο θέμα του φορολογικού ανταγωνισμού που τον χαρακτηρίζεται αρνητικό και επισημαίνεται ότι τέτοιου είδους αρνητικός ανταγωνισμός θα πρέπει να περιστεί κυρίως σε θέματα φορολογικά. Να πω λοιπόν το εξής. Κάποια κράτη-μέλη αν εισήγαγαν την ψηφιακή φορολογία, κατά την άποψή σας, αυτό που θα οδηγούσε, θα στήριζε ή θα μείωνε τον φορολογικό ανταγωνισμό. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Και το δεύτερο, πιστεύετε εσείς ε, ότι ένας ε, ενιαίος, μια ενιαία ψηφιακή φορολόγηση θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη ανάπτυξη και εμβάθυνση των ε, προσφερόμενων υπηρεσιών ή θα αποτελούσε εμπόδιο στο να ακολουθήσουμε αυτή την εξέλιξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας. Η ψηφιακή ε, φορολόγηση είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Οι άνθρωποι μιλάνε πάρα πολύ για το θέμα αυτό. Θα ήταν λοιπόν καλύτερα, κατά την άποψή μου, να προχωρήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι σε εθνικό επίπεδο. Η καλύτερη λύση θα ήταν, όπως ήδη είπα και προηγουμένως, ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε από αυτό το θέμα σε διεθνές επίπεδο, αλλά αν τελικά ακολουθηθεί εθνική λύση, θα μπορούσαν, ή στην περίπτωση αυτή, θα προέκυπταν πάρα πολλές λύσεις. Εμείς στηρίζουμε την ενιαία αγορά των προσφερόμενων υπηρεσιών, ως εκ τούτου ενιαία ψηφιακή φορολόγηση για μας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Πολύ ωραία. Μια χαρά τα πάμε με το χρόνο. Από το ECR, Γιουρίτσα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Θα μιλήσω σλοβακικά. Κύριε Υπουργέ, έχω τρεις ερωτήσεις. όσον αφορά τις προτεραιότητες της Φιλανδικής Προεδρίας. Αφενός μεν, οι δημοσιονομικοί κανόνες δεν τηρούνται πλήρως και γι' αυτό μιλάμε για μεγαλύτερη ευελιξία το οποίο μπορεί να επιτρέπει και στο δημόσιο χρέος να αυξάνεται. Η Φινλανδία μιλάει για την απλούστευση. Αυτό θα μπορούσαμε ε, να το εκλάβουμε ως πιο αυστηρή στάση. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι αν θα προσπαθήσετε να, μειωθούν τα, να μειωθεί το δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη. Ε, δεύτερη ερώτηση. Ε, μια ερώτηση που έχει σχέση με αυτό που συζητήσαμε και με την κυρία Λαγκάρντ. Ε, το ισοζύγιο της ΕΚΤ αυξήθηκε, εκατονταπλασιάστηκε τα τελευταία χρόνια. Και αυτό έχει κάποιες ανεπιθύμητες ανέργειες ε, στην πολιτική των τιμών. Πώς βλέπετε εσείς αυτές τις παρενέργειες αυτής της ε, φιλελευθεροποίησης. Και όσον αφορά την πολιτική για το κλίμα, πιστεύετε ότι οι οικονομικές αναλύσεις συνδέονται με σωστό τρόπο με αυτά τα περιβαλλοντικά θέματα ή χρειαζόμαστε μεγαλύτερο βάθος αναλύσεων. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, η δημοσιονομική πολιτική και ρύθμιση και εναλλακτικέ στο σύμφωνο σταθερότητας. Αυτό με ρωτάτε. Εμεί θέλουμε περισσότερη διαφάνεια και περισσότερο άνοιγμα. Στόχος είναι η ανάπτυξη της νομισματικής πολιτικής να ενισχυθεί και να βελτιωθεί η αξιοπιστία. Είναι πολύ σημαντικό να βελτιωθεί η σταθερότητα, η προβλεψιμότητα ε, του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και γι' αυτό θα πρέπει να αποφύγουμε τη σημερινή περιπλοκότητα. Το Σύμφωνο Ανάπτυξης και Σταθερότητας πρέπει να ε, προσαρμόζεται ε, σε διάφορες οικονομικές συγκυρίες. Θα συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα στο άτυπο ΕΚΟΦΗΝ γι' αυτά. Όσον αφορά τώρα τον ε, απολογισμό ΕΚΤ, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εδώ δεν μπορώ από τη δικιά μου ε, την ιδιότητα να σας απαντήσω σε αυτό. Και η τελευταία σας ερώτηση είχε να κάνει με το περιβάλλον. Κατά πόσο πρέπει να ενσωματώνεται πλήρως στην οικονομία. Κατά τη γνώμη μου, ναι, απολύτως. Κατά τη γνώμη μου, αυτό το οποίο θα ήταν καλό, θα ήταν το ΕΚΟΦΗΝ έχει μία περιβαλλοντική συμμαχία. Και αυτό ακριβώς είναι ε, το οποίο προσπαθώ να κάνω με τον ε, Φιλίνο συναδελφό μου. Είναι πολύ σημαντικό για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Σας ευχαριστούμε. Επόμενος ο μιλητής για ερώτηση, ο Δημήτρης Παπαδημούλης από την ΚΟΕ. Παρακαλώ και έτσι θα κλείσει ο πρώτος γύρος ερωτήσεων. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Αναλαμβάνεται την Προεδρία σε μια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Οικονομία βρίσκεται σε, μπροστά σε μεγάλες ε, προκλήσεις. Γιατί επιβραδύνεται η πορεία της οικονομίας σε αρκετές χώρες, με πρώτη τη Γερμανία, γιατί υπάρχει μπροστά ο κίνδυνος μιας νέας παγκόσμιας ύφεσης και την ίδια ώρα ενώ στους στόχους σας θέτετε την κοινωνική συνοχή και συμμετοχή, το Socially Inclusive EU, όπως αναφέρετε στους γραπτούς σας στόχους, και μιλάτε και για βιώσιμη ανάπτυξη κτλ. Ε, δεν έχουμε ακόμη απαντήσεις από την πλευρά του Συμβουλίου στον προϋπολογισμό, όπου μια σειρά χώρες ζητούν και τις περικοπή κονδυλίων από την πρόταση της Κομισιόν για την κοινή αγροτική πολιτική, την πολιτική συνοχής. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς θα επιτευχθούν όλοι αυτοί οι στόχοι για συνοχή, για συμμετοχική ανάπτυξη της οικονομίας, για αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής με έναν περικεκομένο προϋπολογισμό. Και ένα δεύτερο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Λιντήλα, είναι για την ολοκλήρωση τραπεζικής ενοποίησης. Η Κομισιόν το έχει προτείνει εδώ και χρόνια, το υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι πρέπει να ολοκληρωθεί ο τρίτος πυλώνας της τραπεζικής ενοποίησης με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύης Καταθέσεων, το περίφημο EDIS, το οποίο εκκρεμεί για περίπου πέντε χρόνια. Επειδή η Φιλανδία, αν δεν κάνω λάθος, είναι στις χώρες που στο Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις στο να προχωρήσει η ολοκλήρωση τραπεζική ενοποίησης. Θα ήθελα να σας πω, αν σκοπεύετε σε αυτό το θέμα, να συμβάλλετε θετικά ως Φιλανδική Προεδρία ή θα συνεχίσουμε να παραπέμπουμε το θέμα στις καλέντες. Ευχαριστώ. Kiitoksia Ευχαριστούμε. Ουσιαστικά, οι ερωτήσεις, οι νομισματικές και δημοσιονομικές εξετάζονται από το ΕΚΟΦΗΝ. Αλλά τα θέματα, τα πιο ουσιώδη, τα εξετάζει το Συμβούλιο. Η Φιλανδική Προεδρία προσπαθεί να υποβάλει μια πρόταση και έχουμε δεσμευτεί να προωθήσουμε την υπόθεση. Βέβαια, το timing, το χρονοδιάγραμμα θα αποφασιστεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οπότε είναι πολύ δύσκολο, θα ήταν πολύ τολμηρό να προσπαθήσει κανείς να προβλέψει πότε θα έχουμε αποτελέσματα. Όταν το Συμβούλιο θα πάρει την εντολή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τότε και εμείς θα δράσουμε προκειμένου να καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη λύση και να έχουμε στα χέρια μας κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να συμφιλιώσουμε όλες τις πλευρές και όλα τα συμφέροντα. Τώρα για την Τραπεζική Ένωση. Έχουμε δεσμευτεί να συνεχίσουμε το τεχνικό έργο για την ενίσχυση της Τραπεζικής Ένωσης. Συνεπώς, περιμένουμε για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Και όσον αφορά τις εγγύησεις, εδώ σκοπεύουμε να προχωρήσουμε τις διαπραγματεύσεις για να καταλήξουμε σε λύσεις. Αυτή είναι η πρόθεσή μας. Έχει ξεκινήσει η δουλειά αλλά δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα περίπλοκο το θέμα, χρειαζόμαστε χρόνο για να πετύχουμε. Ελπίζουμε πάντως ότι δεν θα καθυστερήσουν οι διαπραγματεύσεις οι οποίες ε, πρέπει να γίνουν για τις ε, δευτερογενείς αγορές. Thank you. So we ε, Περνάμε στο δεύτερο γύρο. Στέφαν Μπέργκερ, ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Ε, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν πολλές ε, και διαφορετικές εξελίξεις στα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε ότι πολλά κράτη βρίσκονται σε μια τελείως ε, διαφορετική δημοσιονομική, οικονομική, πολιτική κατάσταση και εσείς ο ίδιος είπατε ότι το σύμφωνο σταθερότητας θα πρέπει να προσαρμοστεί. Μήπως μπορείτε λιγάκι να το διευκρινίσετε αυτό, πώς θα μπορέσουμε δηλαδή το χρέος σε ορισμένα κράτη, να το ελέγξουμε καλύτερα, έχοντας επίσης ε, κατά νου ότι η ε, γενικότερη οικονομική κατάσταση τίνει λιγάκι προς ε, την ύφεση. Κατόπιν μιλήσατε για την, τον, την ψηφιακή φορολόγηση και πρέπει να σας πω, δεν το έχω καταλάβει ακόμα καλά, τι θέλετε, έναν τέτοιο ε, φόρο που θα ισχύει σε ολόκληρη την Ευρώπη ή ένας φόρος για κάθε ξεχωριστό κράτος μέλο. Ίσως μπορείτε λιγάκι να το διευκρινίσετε αυτό. Ε, και το τρίτο θέμα που θέλω να δείξω είναι ότι ε, θα θέλαμε να γνωρίζουμε στον τομέα της ψηφιοποίησης θα κρυθούν πάρα πολλά θέματα και είναι επίσης σαφές ότι η οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μια κοινωνία ε, κρίνεται και από τις επενδύσεις που γίνονται στο χώρο της ε, ψηφιοποίησης. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω, στο ΕΚΟΦΗΝ το σκέφτεστε αυτό, το να κάνετε επενδύσεις στον τομέα της ε, ψηφιοποίησης και μάλιστα να πλουστευτούν ε, τα διαδικασίες, δηλαδή να βελτιωθούν οι διαδικασίες παραγραφής ή να δοθούν ίσως κάποια φορολογικά κίνητρα. Ε, αυτές είναι οι ερωτήσεις που θέλω να σας κάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Σύμφωνο Σταθερότητας, κοιτάξτε, ήδη είπα σχετικά με αυτό το σύμφωνο ότι ε, έχουμε κατά νου διάφορες εναλλακτικέ λύσεις για να βελτιώσουμε την προβλεψιμότητα, την διαφάνεια και ο στόχος είναι να ισχυθεί το ε, πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να γίνει και πιο αξιόπιστο. Όσον αφορά την ψηφιακή φορολόγηση, ο στόχος ε, είναι να ε, έχουμε μία εναρμόνιση. Βεβαίως δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει σε διεθνές επίπεδο. Να έχουμε εθνική φορολόγηση, αλλά να είναι εναρμονισμένη αυτή η εθνική φορολόγηση. Τώρα, όσον αφορά τις ψηφιακέ επενδύσεις στο ΕΚΟΦΗΝ, να σας πω ότι δεν το συζητήσαμε καθόλου το θέμα αυτό. Ο κύριος Μαυρίδης, παρακαλώ, για τους σοσιαλδημοκράτες. Θα είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένος, ε, γιατί οι ερωτήσει μου είναι πολύ συγκεκριμένε και θέλω συγκεκριμένες απαντήσεις. Μήπως μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς σημαίνει ε, βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη, κυρίως σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση μου είναι η εξής. Ο κύριος Παπαδημούλης έκανε μια ερώτηση, ε, συνεχίζω με την ίδια, προς την ίδια κατεύθυνση και θέλω να σας πω ότι δεν αφορά εσάς αυτό που θα πω, αλλά γενικότερα η εφαρμογή του τρίτου πυλώνα της ε, Τραπεζικής Ένωσης δεν μας πείθει. Και να σας πω γιατί βρίσκομαι εδώ ε, πέντε χρόνια, ήμουν εδώ καθ' όλη την προηγούμενη θητεία και ε, κατά την άποψή μου η αντίσταση προς την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης δεν ήταν τόσο τα τεχνικά στοιχεία, η παρεμφερή, που αυτό θα το κατανοούσαμε. Η αντίδραση ήταν περισσότερο πολιτικής φύσεως. Και το δικό μου το ερώτημα είναι το εξής. Λαμβάζον, λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αρχική σας παρέμβαση είπατε ότι η προτεραιότητά σας είναι η ανταγωνιστικότητα και η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μπορείτε μήπως να μας εξηγήσετε γιατί δεν υπάρχει ε, πρόοδος στην Τραπεζική Ένωση. Πώς μπορούμε να μιλάμε για CMU χωρίς ε, την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Γιατί αν δεν προχωρήσουμε, ακόμα και μετά από κάποια χρόνια θα βρισκόμαστε εδώ και θα διαμαρτυρόμαστε για τον τρίτο πυλώνα, ενώ αρκετά κράτη-μέλη θα υποφέρουν από ε, κοινωνικά και οικονομικά και άλλα προβλήματα, ακριβώς γιατί δεν εφαρμόζονται οι δύο πρώτοι πυλώνες. Το θέμα δεν είναι μόνο η πολιτική, το θέμα είναι ηθικής φύσεως και εμεί έτσι κατανοούμε κοινέ αξίες και κοινή μοίρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα παρακαλώ ή δυνατόν να σχολιάσετε ακριβώς αυτά που σας είπα. Σας ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά ε, τη βιώσιμη χρηματοδότηση, ο στόχος είναι οι, οι οικονομικές ε, χρηματοπιστωτικές αγορές να στηρίξουν τη μετάβαση προς μια πιο πράσινη οικονομία. Ε, τι ακριβώς τώρα σημαίνει πράσινη οικονομία. Είναι βέβαια ένας ορισμός όπου το βασικότερο είναι οι ενέργειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή σε όλο τον κόσμο είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας. Και όσον αφορά το Eurogroup, ε, εργαζόμεθα για την ολοκλήρωση της ε, Τραπεζικής Ένωσης. Και εδώ ε, θέλουμε να έχουμε ένα πρόγραμμα εξασφάλισης των καταθέσεων, αλλά αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, δεν θα έχουμε χρόνο να το πράξουμε εμείς στην Προεδρία μας, αλλά είμαι αδιαμφισβήτητα υπέρ της ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης. Λουίζα Πόρη, την επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, που ήρθατε στην Επιτροπή μας σήμερα. Θα σας ζητήσω να μας σχολιάσετε το Brexit, γιατί ζούμε σε ταραγμένες εποχές και η χώρα μου, το Ηνωμένο Βασίλειο, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο αυτών των δυσκολιών στην Ευρώπη. Όπως και άλλοι ε, φίλοι Ευρωπαίοι, θα ήθελα να αποφύγουμε ένα καταστροφικό Brexit χωρίς συμφωνία που θα ήταν εις όλων των οικονομιών μας. Θα προτιμούσα να μην έχουμε καν το Brexit η στενή οικονομική συνεργασία μας έχει ωφελήσει όλους. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω καταρχήν, ποια, πείτε μας ποια βήματα έχουν ληφθεί σε επίπεδο Συμβουλίου για να μετριαστεί ο αντίκτυπος σε περίπτωση ξαφνικής εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, και αυτό είναι σημαντικό για μα που πιστεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τι οικονομικέ ανισορροπίες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίω στην Ευρωζώνη που έχουν τροφοδοτήσει τα επιχειρήματα των λαϊκιστών που υπονομεύουν τώρα ακόμη και την ύπαρξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά την ανεργία των νέων, η αντιμετώπιση τη κρίση στην Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία ε, και η στασιμότητα από την οικονομική κρίση δεν έχουν βοηθήσει στα, στην επιχειρηματολογία μας. Στο πλαίσιο αυτό, οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις ε, τις οποίες έχετε κατά νου είναι κέρια σημασίας ε, για την προστασία της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Είναι πολύ επίκαιρο το ερώτημά σας. Δυστυχώς ε, δεν είναι αντικείμενο των αρμοδιοτήτων μου ως Προεδρεύοντος του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ. Όπως γνωρίζετε, η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα αυτό είναι σαφής έχουμε μια συμφωνία για τον Brexit και δεν ξανανοίγουμε αυτή τη συμφωνία που έχει ήδη κλείσει. Το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ ε, καταβάλει προσπάθειες ε, προς την κατεύθυνση του να λειτουργούν οι αγορές παραγόγων και στην περίπτωση μιας εξόδου χωρίς συμφωνία. Σχετικά με το γενικότερο ερώτημα που θέσατε για τη φιλελεύθερη δημοκρατία είναι έργο όλων των πολιτικών ε, να διασφαλίσουν ε, τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Όλοι πρέπει να έχουν τη συλλογική ευθύνη για τη διατήρηση της δημοκρατίας. Νομίζω ότι έγινε και μια ερώτηση για τις ανισορροπίες στην Ευρωζώνη. Αυτό είναι κάτι στο πλαίσιο του ΕΚΟΦΗΝ, πώς μπορείτε να σχολιάσετε από αυτού. Niin, herra puheenjohtaja. Itse asiassa Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτές οι εσωτερικές ανισορροπίες είναι αντικείμενο του Eurogroup και όχι του ECOFIN. Εξάλλου είμαι και εγώ ίδιος ε, νέο μέλος, οπότε δεν έχω να σας δώσω κάποια απάντηση από αυτού. Τζέσικα Πολφιέρ, εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Λεντιλέ για την παρουσίασή σας. Βλέπουμε την επιβράδυνση της οικονομίας στην Ευρώπη, βλέπουμε τις προβλέψεις, βλέπουμε ενδεχόμενα όπως το Brexit και οι εμπορικές διαμάχες. Αυτά μπορεί να είναι ακόμη πιο επιζήμια για την ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι ε, θεμελιώδου σημασία να χρησιμοποιούν τα κράτη-μέλη τι ευκαιρίε που δίνονται από την οικονομική ανάπτυξη για να εφαρμόσουν τι απαραίτητε μεταρρυθμίσει εγκαίρω, πριν έρθουν οι χειρότερε εποχέ. Θα ήθελα να σα ρωτήσω λοιπόν πώς θα ενθαρρύνει η Προεδρία σας τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τις αναχώρα συστάσει, ιδιαίτερα για το δημοσιονομικό έλλειμμα, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ύφεση ε, με ε, αυξανόμενες τιμές ε, ε, ε, αποδόσεις ομολόγων. Μερικές τέτοιες συστάσεις δεν έχουν εφαρμοστεί, μερικές φορές και καθόλου. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Η σταθερότητα και η ανάπτυξη είναι αντικείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δικό μας καθήκον είναι να προωθούμε τις εργασίες του Συμβουλίου στους τομείς αυτούς. Ελπίζω ότι όλα τα κράτη-μέλη θα ακολουθούν αυτές τις προτάσεις και το πλαίσιο που τίθεται. Επόμενος, Άλφρετ Σάντ, Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις και την καθεμία θα συνοδεύει και μια ερώτηση. Πρώτον, το ευρωπαϊκό οικονομικό σενάριο είναι χαμηλός πληθωρισμός, ενώ η νομισματική πολιτική εφαρμόζεται για να ε, πετύχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει μια τεράστια περίοδος χαμηλής ανάπτυξης και έχουμε τώρα μπροστά μας έναν εμπορικό πόλεμο Ηνωμένων Πολιτείων Κίνας. έχουμε μία πολιτική που ακολουθούμε, η οποία ε, όμως έχει εφαρμοστεί και πριν από 40 χρόνια στην Ευρώπη, ενώ η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Η κατάσταση τότε δεν έχει κανένα νόημα σήμερα. Δεσμεύονται οι χώρες μας πολύ περισσότερο από ό,τι δεσμεύονται αντίστοιχα Ηνωμένε Πολιτείες, Κάτι το οποίο φυσικά μας κοστίζει. Δεν έχει νόημα κάτι τέτοιο η προσέγγιση μας βασίζεται σε μεσοπρόθεσμες ε, προσδοκίες. Οπότε ρωτάω, δεν ήρθε η ώρα για να αλλάξουμε μοντέλο. Δεύτερον, η διαχείριση των διαφόρων holdings. Σε περιπτώσεις ε, έκτακτες έχουμε διαχειρίσει που βασίζεται σε πληρωμές. Όμως η δημιουργία των, του, του χρήματος έχει επιτραπεί τελευταία. Η πρόταση τώρα του Facebook έχει να κάνει με εκατομμύρια πελάτες για ένα νέο νόμισμα. Και μάλιστα τώρα που υπάρχει και το Brexit πώς θα αντιμετωπιστεί από τις αρχές. Η σύγκρουση συμφερόντων με αυτά που προτείνονται είναι σαφής. Δεν ξέρουμε βέβαια πώς ακριβώς θα λειτουργήσει το σύστημα, αλλά σίγουρα η κυριότητα του δικού μας τραπεζικού συστήματος θα πληγεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν μέχρι τώρα πάντα πάρα πολύ προσεκτική. Εσείς τι άποψη έχετε? Έχει τεθεί καθόλου το θέμα? Ευχαριστώ. Για αυτές τις τοποθετήσεις σας και για τις ερωτήσεις. Όπως είπα και νωρίτερα, εξετάζουμε εναλλακτικέ για να βελτιώσουμε την προβλεψιμότητα και την ε, διαφάνεια στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί το πλαίσιο ε, της πολιτικής μας και να βελτιωθεί και η αξιοπιστία της. Εγώ δεν νομίζω ότι, για παράδειγμα, σε έξι μήνες προεδρίας μπορούμε να πετύχουμε σημαντική πρόοδο. Η συζήτηση για τα κρυπτονομίσματα. Ε, συζητήθηκε το θέμα με τους κυβερνήτες, συγγνώμη, με τους διοικητές των ε, κεντρικών τραπεζών και η συζήτηση αυτή θα συνεχιστεί και στο ΕΚΟΦΗΝ. Προς το παρόν δεν την έχει συζητήσει αυτή την υπόθεση στο ΕΚΟΦΗΝ. Ε, το επόμενο σλότ είναι για τους πράσινους, αλλά οι πράσινοι δεν θέλουν να πάρουν το λόγο από ό,τι έχω καταλάβει. Οπότε, ταυτότητα και δημοκρατία, μπέκ. Πάλι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ στον αγώνα κατά της ε, ε, κατά του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος και της φοροδιαφυγής. Όπως ξέρετε, υπάρχει μια νέα οδηγία για την αντιμετώπιση της παράνομης των εισόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το Μάρτιο του 2019 έγιναν έρευνες και με βάση τα πορίσματα στη Φινλανδία το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος αυτή τη στιγμή επεκτείνεται. Η Φινλανδία, λόγω των πακτικών που ακολουθεί για το άνοιγμα λογαριασμών, δηλαδή η Φινλανδία ζητάει μόνο τον αριθμό ταυτότητας και για να κάνει κανείς χρήση λογαριασμού, για να ανοίξει λογαριασμό, είναι πολύ ελκυστική αυτή η χώρα. Ως εκ τούτου, τον Μάρτιο του 2019, η Φινλανδία όρισε έναν ε, θεματοφύλακα που ελέγχει τα θέματα του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, αλλά με βάση μια έκθεση που έγινε στην Φινλανδία διαπιστώθηκε το 2009, την άνοιξη του 2019, ότι στη Φινλανδία υπάρχουν πάρα πολλοί ε, που πρέπει όμως να έχουν ειδικέ γνώσεις για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Και γι' αυτό λοιπόν σας ερωτώ, πιστεύετε εσείς ότι η Φινλανδία όσον αφορά την νομιμοποίηση παράνομων εσόδων από παράνομες δραστηριότητε υστερεί η Φινλανδία σε σχέση με άλλες χώρες. Και αν ναι, ε, τι πιστεύετε, τι πρέπει να μάθει η Φινλανδία και πού ακριβώς πρέπει απαρέγκλητα και απαραίτητα να βελτιωθεί. Θα σας απαντήσω. Φροντίζουμε για την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού νομοποίησης χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες. Υπάρχει το ΕΦΑΤΕΦ που ερευνεί το θέμα και έχουν γίνει συστάσεις από τον οργανισμό αυτό που εφαρμόζονται μάλιστα σήμερα για το θέμα του ξεπλήματος χρήματος. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύθηκε το 2018 όταν τροποποιήθηκε η οδηγία η σχετική με την ε, νομιμοποίηση παράνομου χρήματος. Ευχαριστούμε. Τσέσικα Στέγκαρτ από το ECR παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αξιότιμε Υπουργέ. Ανακοινώσατε πρόσφατα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Φιλανδία εξετάζουν τη δυνατότητα να απαγορεύσουν τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία. Έχω εμπειρία 25 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και ξέρω ότι οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται βάσει γεγονότων και οι έρευνες δείχνουν ότι θέλουμε να αποκτήσουμε αρρώσιμη γη και ότι έχουν μειωθεί κατά 25% οι σχετικές ε, γης και υπάρχει και αύξηση στα δάση τα τελευταία 25 χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που προτείνεται θέτει σε κίνδυνο την παρετέρω ανάπτυξη ακόμα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν πραγματικά σας ενδιαφέρει η ανάπτυξη και οι πυρκαγιές στον Αμαζόνιο, τότε δεν πιστεύετε ότι το μέτρο που προτείνετε θα είναι αντιπαραγωγικό. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Αυτό που είπα εγώ είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να μελετήσει το θέμα των εξαγωγών βοήου κρέατος από την Βραζιλία σε εμά. Το πιο σημαντικό τότε ήταν το θέμα των πυρκαγιών που δεν αφορούν μόνο τη Βραζιλία και που θα έπρεπε να απασχολήσουν την Επιτροπή. Οπότε πρέπει να βρούμε λύσεις οι οποίες να λειτουργούν και οι οποίες έχουν να κάνουν με την οικονομία. Όπως για παράδειγμα υπάρχει δυνατότητα βάσει μιας παρουσίασης, μιας πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα. Προς το παρόν όμως δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Πολύ ωραία. Τώρα στη διαδικασία ΚΑΤΣΙΑ, κυρία Μαργαρίτ Μαγκές. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας δώσατε ε, και επίσης ε, και για όλα τα άλλα που είπατε. Πρώτα απ' όλα, σχετικά με το Brexit, ε, λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις που δώσατε στο Brexit, έχω μόνο μία ερώτηση, την άλλη την απαντήσατε, αλλά προκύπτουν βέβαια και άλλες ερωτήσεις σε σχέση με την πρόοδο που σημειώνει η διαδικασία Brexit. Να πω λοιπόν το εξής, στην Επιτροπή προϋπολογισμών δεν ε, είχαμε κανένα εκπρόσωπο της Προεδρίας. Μέχρι τώρα δεν μας έκανε την τιμή. Ε, αυτό βέβαια ίσως να έχει περισσότερο σχέση με τον προϋπολογισμό και όχι με την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Ερωτώ. η Φινλανδική Προεδρία προτίθεται να διεκδικήσει συμφωνία επί του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου κατά τη διάρκεια αυτού του εξαμήνου. Και δεύτερο ερώτημα αφορά στην Ευρωζώνη, στην πρόταση η Κομισιόν να παρουσιάσει ένα μηχανισμό που θα είναι το σημείο εκκίνησης για την ε, σύσταση ε, προϋπολογισμού της Ευρωζώνης. Ποια ακριβώς είναι η θέση της ε, Φινλανδικής ε, Προεδρίας. Τι προτίθεστε να προτείνετε σε αυτόν τον τομέα. Καταρχήν, όσον αφορά στην κατάρτιση προϋπολογισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεύτερον όσον αφορά στα ποσά που θα προταθούν. Ως πρόεδρος του ΕΚΟΦΗΝ πιστεύετε εσείς ότι το ποσό που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ικανοποιητικό για να υπάρχει μια δημοσιονομική ικανότητα στην Ευρωζώνη. Ευχαριστώ πολύ Δυστυχώς πρέπει να σας πω δεν ξέρω γιατί δεν πήγε ακόμα κανένας εκπρόσωπος της Φινλανδικής Προεδρίας στην ε, Επιτροπή Προεπλογισμών, παρότι εκεί υπάρχει μέλος από την ε, Φινλανδία. Όσον αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, αυτά τα θέματα συζητιούνται κυρίως στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εγώ προσωπικά ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια της Φινλανδικής Προεδρίας θα μπορέσουμε να σας καταθέσουμε μια εικονοποιητική πρόταση ε, και τέλος ε, θέλω να σας πω ότι ο χρόνος ε, καθορίζεται από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η Φινλανδία θα συνεχίσει αυτή τη δουλειά και με βάση τις αποφάσεις του Eurogroup. Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι ο προϋπολογισμός της Ευρωζώνης. Έχουμε λοιπόν ξεκινήσει τη νομοθετική εργασία τουλάχιστον όσον αφορά το πρόγραμμα στήριξης των μεταρρυθμίσεων. Το ΕΚΟΦΗΝ εξακολουθεί να συζητά κάποια θέματα που εκκρεμούν. Είμαστε σε επαφή με τον πρόεδρο του Eurogroup όσον αφορά σε αυτά τα ερωτήματα. Και όσον αφορά στο ποσό του ε, προπολογισμού ε, δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο ποσό να αναφέρω. Ε, δεν μπορώ να σχολιάσω οτιδήποτε. Κύριο Νικολάου. Κύριε Υπουργέ, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες σχεδιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και εφαρμόστηκε ε, με τη συμφωνία των κυβερνήσεων σε αυτές τις χώρες μια σκληρή αντιλαϊκή πολιτική ε, μπροστά στην καταπολέμηση της κρίσης και της ύφεση. Ήταν μια πολιτική η οποία εστίασε στη θωράκιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε περίοδο καπιταλιστικής κρίσης, με μέτρα ενίσχυσης της κερδοφορίας των καπιταλιστικών ομήλων, με ανακεφαλαιοποιήσεις και ενέσεις ρευστότητα στις τράπεζες, μια ρευστότητα όμως η οποία προήλθε από το τσάκισμα των μισθών, των συντάξεων, των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Παρά τη φιλολογία ότι τα δύσκολα τώρα έχουν περάσει, η παρούσα οικονομική κατάσταση διεθνώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει το αντίθετο. Εξάλλου, τα μνημόνια είναι δέσμοι μέτρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήρθαν για να μείνουν. Αυτό φαίνεται από τη συζήτηση που ανοίγει σήμερα για το λεγόμενο δημοσιονομικό χώρο που μεταφράζεται σε μεγαλύτερο έδαφο για την κερδοφορία των μεγάλων ομήλων. Επανέρχονται αυτά τα ζητήματα πιο έντονα με επίκεντρο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, εστιάζοντα όχι στι τεράστιε οφειλέ που έχουν οι επιχειρηματίε και επιχειρήσει, αλλά στου εκατοντάδε χιλιάδε μικροφιλέτε σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Χιλιάδες απολύσεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα μαζί με την έναρξη εκαθάρισης κόκκινων δανείων από ιδιωτικά funds, κατασχέσεις καταθέσεων, 120.000 πληστηριασμοί στην Ελλάδα, οι οποίοι ξεκινούν από σήμερα 4 Σεπτεμβρίου με το ηλεκτρονικό σύστημα. Θα ήθελα να απαντήσετε αν μπορείτε πώς τοποθετήσετε στο αίτημα που υπάρχει για την ομοθετική απαγόρευση πληστηριασμών των λαϊκών κατοικιών και την ομοθετική απαγόρευση Κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών μισθοδοσίας και συντάξεων από το κράτος, τι τράπεζε ή τα ιδιωτικά funds. Ευχαριστώ. Kiitoksia kysymyksestä. Σα ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά στους ε, αναγκαστικούς ε, πληστηριασμούς ε, και στην κατάσχεση των συντάξεων. Σας πω κάτι, αυτό δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΕΚΟΦΗΝ. Είναι περισσότερο εθνικές αποφάσεις που λαμβάνονται από τα κράτη-μέλη. Ε, τα μέτρα σταθεροποίησης και εξυγίανσης δεν αποφασίζονται από το ΕΚΟΦΗΝ, αλλά από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Κατανοώ πάντως τις ανησυχίες σας και ελπίζω ότι σε συνεργασία με την καινούργια κυβέρνηση θα μπορείτε να ε, λάβετε μέτρα έτσι ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση θέση των Ελλήνων πολιτών. Ο κύριος Φουγκοσάνκ από τους Σοσιαλδημοκράτες. Εδώ, αριστερά. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ για τη συζήτηση που κάναμε μέχρι τώρα, γιατί ασχοληθήκαμε με πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Έχω ένα αρκετά ευρύ ερώτημα το θέμα της αύξησης των ανισοτήτων που διαπιστώνουμε. Διαβρύνονται οι ανισότητες μεταξύ φτωχών και πλουσίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Αυτή η τάση προς την ανισότητα αποτελεί μια αδικία όσο τη βλέπουμε εμείς ε, ως ομάδα σοσιαλιστών και δημοκρατών και αν συνεχιστεί θα αποτελεί και απειλή για την οικονομική σταθερότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζητήσατε πολλά και ποικίλα θέματα. Τραπεζική Ένωση, ρυθμίσεις ε, στον φορολογικό τομέα, φορολογικούς παραδείσους, ε, πολιτικές λιτότητας. Πιστεύετε ότι είναι πρόβλημα και η αύξηση των ανισοτήτων. Πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση και συμφωνείτε ότι ίσως και η, Ευρωπαϊκή, και η ε, Φινλανδική Προεδρία μπορεί να κάνει κάτι τι πιστεύετε ότι είναι το πιο σημαντικό το οποίο θα μπορούσε να κάνει η Φιλανδική Προεδρία ή που θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε για να αλλάξουμε αυτή την τάση αύξησης των ανισοτήτων. Ευχαριστώ. Όπως είπατε και εσείς, είναι ένα ευρύτατο θέμα, με τεράστια σημασία βέβαια. οι ανισότητες και οι κοινωνικές ανισότητες όντως αυξάνονται σε πολλές χώρες. Ο καλύτερος τρόπος για τη βελτίωση και για να επιτύχουμε μια ισορροπημένη κατάσταση είναι να επιδιώξουμε να έχουν θέσεις εργασίας οι πολίτες ώστε να μπορούν να κερδίζουν τη ζωή τους. Και η ανάπτυξη είναι ένας από τους τρόπους για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των αυξανόμενων ανισοτήτων. Κατά την Φινλανδική Προεδρία έχουμε θέσει ως προτεραιότητα το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και η κοινωνική ανισότητα και η κλιματική αλλαγή ε, ε, αποτελούν προτεραιότητές μας. Το θεωρώ και εγώ πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα των ανισοτήτων. Αλλά αυτή τη στιγμή θέσαμε ως προτεραιότητα κυρίως την κλιματική αλλαγή. Ελπίζουμε ότι θα μας βοηθήσει στην ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην αύξηση ε, της ισορροπίας. Ευχαριστώ, κύριε Γκιώρη, από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Χαιρετίζουμε τις πρωτοβουλίες σας για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπό αυτό το πνεύμα υποστηρίζουμε την εμβάθυνση της Νομισματικής Ένωσης και της Τραπεζικής Ένωσης και της περαιτέρω ανάπτυξης των Ένωση της Ένωσης Κεφαλαίου Αγορών. Κάτι που με ανησυχεί και το ίδιο ερώτημα έθεσα και στην κυρία Λαγκάρντ σχετικά με την ειρηνική συνύπαρξη Ευρωζώνης και χωρών εκτός Ευρωζώνης. Σε αυτό το πλαίσιο ε, μπαίνει και ο προϋπολογισμός της Ευρωζώνης που δημιουργεί ανησυχίες στις χώρες εκτός Ευρωζώνης. Έχουμε λίγο πολύ το ίδιο ρυθμιστικό πλαίσιο. Είμαστε στην ίδια ενιαία αγορά και πιστεύουμε ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωζώνης θέτει κάποιους κινδύνους για την αρμονική συνεργασία μεταξύ χωρών Ευρωζώνης και εκτός Ευρωζώνης. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν τη γνώμη σας από ε, αυτού. Ποιο είναι το σχέδιο της Φινλανδικής Προεδρίας για να αντιμετωπίσει Αυτέ τι ανησυχίε των χωρών εκτό Ευρωζώνη και ποια είναι τα σχέδιά σα συγκεκριμένα για τον προπολογισμό τη Ευρωζώνη. Ευχαριστώ. Kiitoksia. Kiitoksia kysymyksestä. Merkittävä kysymys ja on ollut keskustelu. Σας ευχαριστώ και αυτή η ερώτηση είναι πολύ σημαντική. Το έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό ήδη σε προηγούμενες ερωτήσεις. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή έχει ως εξή. Έχουμε κάνει διαβουλεύσεις με χώρες εκτός Ευρωζώνης και μετά από τις διαβουλεύσεις αυτές θα πρέπει να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα και να αξιολογήσουμε τι θα γίνει περαιτέρω. πώς θα μπορέσουμε ε, να βοηθήσουμε ε, στην εξομάλυνση των πιθανών προβλημάτων. Ε. Ωραία. Δεν υπάρχει κανένα άλλο στη διαδικασία ΚΑΤΣΔΙ. Αγαπητέ Υπουργέ, μήπως θέλετε να πείτε κάτι για να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Όχι, ωραία. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να ξέρετε ότι μπορείτε να βασίζεστε στη δική μας συνεργασία. Ελπίζω να ξανασυζητήσουμε αυτά τα θέματα στο μέλλον. Τώρα, έξι λεπτά διακοπή και θα περάσουμε στην επόμενη ακρόαση. Thank you. Thank you So, dear colleagues, let me, let me start. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Είναι η τέταρτη ακρόαση μας για σήμερα. Είναι η πιο σύντομη έτσι έχουμε προβλέψει. Πρόκειται για το διορισμό αντιπροέδρου του Υποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στις 11 Φεβρουαρίου η κυρία Λάμπερ Σάκιον που είναι η αντιπρόεδρος έληξε η εντολή της και ενημερωθήκαμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε τον κύριο Μέρς να οριστεί αντιπρόεδρος ως μέλος εκτελεστικής επιτροπής είναι μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου της επόμενης χρονιάς. Η διαδικασία βασίζεται στο άρθρο 26.3 του κανονισμού του SSM που λέει ότι επιλέγεται ο Αντιπρόεδρος από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής ε, Τράπεζας. Η ακρόση που έχουμε σήμερα είναι πολύ σημαντική, να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει επικοινωνία μεταξύ μας. Εσείς ε, λοιπόν τώρα θα έχετε το λόγο για πέντε λεπτά εισαγωγικά και μετά θα ακολουθήσουν ερωτήσεις. Πέντε λεπτά η καθεμία μαζί με την απάντηση. Οπότε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον συνάδελφο από την Κεντρική Τράπεζα. Θέλω να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι και πάλι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή τη φορά έρχομαι για να σας εξηγήσω γιατί το Διευθυντικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πρότεινε να αναλάβω ε, εγώ να περάσω πρώτα από έλεγχο και να αναλάβω εγώ τα εποπτικά αυτά καθήκοντα. Όταν δημιουργήθηκε ο SSM, εγώ ήμουν επικεφαλής στην προετοιμασία του εποπτικού αυτού μηχανισμού. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο δεν γνωρίζω. Προηγουμένως, σε εθνικό επίπεδο ήμουν διοικητής της Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας και εκεί είχα αναλάβει την εποπτεία για ο καιρό εκ μέρους Εθνικής Κεντρικής Τράπεζας. Επίσης ήμουνα στο Διοικητικό Συμβούλιο τοπικών ε, εποπτικών αρχών και στο, Υπουργό, στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου και εκεί εργάστηκα και υπό την ιδιότητα αυτή παρακολουθούσα τις εποπτικές δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα πια έχουμε τον SSM τον ενιαίο μηχανισμό και έχει προετοιμαστεί πολύ καλά και εγώ τώρα, εφόσον αναλάβω, θα συνεχίσω το προπαρασκευαστικό αυτό έργο. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ κάπως μαζί σας τρεις διαστάσεις που με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Και εφόσον ε, εγκρίνεται το διορισμό μου, θα φροντίσω να τις υλοποιήσω κιόλα. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε εποπτεία πιο προχωρημένη. Ε, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ό,τι έχει απομείνει από την κρίση και ότι μας κληρονόμησε η κρίση και από το 2014 είδαμε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ότι ήταν η πιο δύσκολη υπόθεση που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Ευτυχώς περίπου 50% έχουν μειωθεί τα δάνεια αυτά και ακούσατε και σήμερα το πρωί τον ε, πρόεδρο που είπε ότι έχει βελτιωθεί σημαντικά η κατάσταση και έχει αυξηθεί και το κεφάλαιο των τραπεζών. Όμως δεν μπορούμε να κοιτάμε μόνο πίσω, πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Σε ένα περιβάλλον λοιπόν αδύναμης προοπτικής ανάπτυξης, δεν ε, μπορούμε να ε, αφήσουμε περιθώριο για νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η εποπτεία λοιπόν είναι αυτή η οποία πρέπει να διασφαλίσει ότι υπάρχουν σωστές προδιαγραφές και σωστές ε, διατάξεις που ισχύουν και τα επιχειρηματικά μοντέλα όταν αλλάζουν να είναι βιώσιμα και ό,τι οι κινδύνου ελοχεύουν να φροντίζουν να αντιμετωπίζονται κατάλληλα. Δεύτερον, διαφάνεια. Ακούσατε σήμερα το πρωί και τον πρόεδρο και τον ρωτήσατε σχετικά. Η διαφάνεια στην εποπτεία είναι κάτι το οποίο προσυπογράφω και εγώ απόλυτα. Γιατί κατά τη γνώμη μου η μακροπροληπτική εποπτεία σημαίνει και δημοκρατική λογοδεσία, γιατί ουσιαστικά προβλέπει τις επιπτώσεις που θα υπάρχουν ε, στα χρήματα των ε, φορολογούμενων σε εθνικό επίπεδο προς το παρόν. Οπότε όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει έχουν γίνει προς την κατεύθυνση του να μειωθεί ακριβώς αυτός ο αντίκτυπος. Η εποπτεία λοιπόν πρέπει να είναι προβλεπόμενη, σαφής και να ενισχύει την διαφάνεια να υπάρχει καλύτερη συνοχή, καλύτερη συγκρισιμότητα όταν έχουμε δηλαδή τα αποτελέσματα των τραπεζών να μπορούμε να τα συγκρίνουμε πιο εύκολα. Και πάλι όλα αυτά επιτρέπουν να υπάρχει μια ισότιμη κατάσταση μεταξύ όλων των ε, ιδρυμάτων τα οποία βρίσκονται υπό εποπτεία καταλαβαίνουμε καλύτερα τους τραπεζικούς κινδύνους και έτσι μπορούμε να προκαταλαμβάνουμε τις δράσεις μας, δράσεις εποπτείας. Πρέπει να υπάρχει βέβαια και πειθαρχία στην αγορά. Πάντως εδώ πρέπει να πω και το εξής. Πρέπει να υπάρχει μια καλή ισορροπία, γιατί ευαίσθητες πληροφορίες πρέπει να ε, παραμένουν απόρριτες, γιατί αλλιώς θέτουν σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Οπότε μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα έχουμε καταλήξει σε συγκεκριμένες προσεγγίσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ μας. Και έτσι έρχομαι τώρα στην τελευταία διάσταση που θα ήθελα να υλοποιήσω. Και αυτή είναι η νομιμότητα των εποπτικών δράσεων. Κατά τη γνώμη μου αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, όταν υπάρχουν ανησυχίες, ότι μπορεί να υπάρχουν εντάσεις ανάμεσα στην νομαστική, νομισματική δράση και την εποπτική δράση, πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Και δεύτερον, και λειτουργικά υπάρχει διάκριση στους τομείς αυτούς ε, πολιτικής ανάμεσα στην νομισματική πολιτική. Υπάρχουν διαφορετικά κτίρια, διαφορετικές συνεδριάσεις, διαφορετικοί στόχοι, αλλά πρέπει να παραδεχτώ παρόλα αυτά ότι αντιμετωπίζουμε νομικές προκλήσεις γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στον εποπτικό κλάδο μας ζητούν να εφαρμόζουμε εθνική νομοθεσία. Η εθνική νομοθεσία όμως δεν έχει ενσωματώσει πλήρως με ομοιόμορφο τρόπο τις ευρωπαϊκές οδηγίες, οπότε μερικές φορές υπάρχει κατακαιρματισμός. Η δεύτερη πτυχή της νομιμότητας είναι ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει και αυτά να σέβονται την εντολή τους και να δρουν στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ή του εθνικού ανάλογα δικαίου. Πρέπει λοιπόν η υποπτική μας δράση να γίνεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ευρωπαϊκής ως επιτοπλίστων. Και αυτά είναι πράγματα τα οποία αποφασίζουν οι συνομοθέτες, δηλαδή το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και από εκεί πέρα υπάρχουν και κάτι άλλα πιο ε, ειδικευμένα θέματα προδιαγραφών που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι ερωτήσεις έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μέρς. Τώρα, πολιτικές ομάδες πρώτα. Πέντε λεπτά. Παρακαλώ, μια που κράτησε λίγο παραπάνω εισαγωγή, αλλά μας βοήθησε πολύ νομίζω για τη συζήτησή μας. Μάρκος Φέμπερ πρώτα απ' όλα, ΕΛΚ. Σε ευχαριστώ πολύ. Ε, σας καλωσορίζουμε που ξανάρχιστε εδώ. Έχετε έρθει αρκετές φορές. Έχω δύο σύντομες ερωτήσεις. Το Νοέμβρη του 2018 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επισήμανε τους μεγάλους κινδύνους που υπάρχουν ε, από την μόχλευση της ε, χρηματοδότησης. Και το 2018 στο πλαίσιο της Financial Stability Reviews και εκεί επισημάνθηκε σχετικά με τον κίνδυνο αυτό από άλλες πλευρές. Ρωτώ λοιπόν ε, ποιοι είναι ακριβώς αυτοί οι κίνδυνοι στην περίπτωση της μόχλευσης, της χρηματοδότησης. Εσείς έχετε κάποια εικόνα για το ε, κατά πόσον ε, ε, το Εποπτικό Ταμείο αντιμετωπίζει και αυτό τέτοιου είδου κινδύνους και υπάρχουν σχετικές οδηγίες για να αντιμετωπιστούν. Το δεύτερο είναι στην ρυθμιστική πρόκληση για αυτή την περίοδο. Μία πρόκληση θα είναι η ολοποίηση της Βασιλείας 3 Πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου ότι οι κεφαλαϊκές απαιτήσει για τις ευρωπαϊκές τράπεζες ε, για τις 26 κιλίους ε, θα αυξηθεί κατά 20%. Τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ε, τα οποία θέλουν την μεγαλύτερη εποπτεία υποφέρουν από τις προδιαγραφές για το περίφημο output flow. Εσείς ε, θεωρείτε ότι οι τράπεζες που εποπτεύονται από το Εποπτικό Ταμείο διατρέχουν κίνδυνο και τι είδους αναλύσεις εξάγεται από αυτό το θέμα σχετικά με την ολοποίηση υλοποίηση της, ε, του πακέτου της Βασιλείας. Um, indeed. Uh, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις ερωτήσεις. Θέλω να σας πω ότι η μόχλευση της χρηματοδότησης είναι ένα από τα θέματα που λαμβάνουμε ιδιαίτερα σοβαρά υπόψη μας. Στον δικό μας τον μηχανισμό, τον SSM, ε, το Εποπτικό Συμβούλιο. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν κίνδυνοι οι οποίοι θα μπορούσαν να απορρεύσουν ε, και από δευτερογενείς επιπτώσεις της συστημικής διάστασης. Αυτά ε, θα μπορούσαν να προκύψουν σε μοχλευμένα δάνεια. Στο Εποπτικό Συμβούλιο ανησυχούμε πάρα πολύ για το ότι καθυστερούν τα default Βεβαίως ε, υπάρχουν συνέπειε από αυτή τη συμπεριφορά και τα αυξανόμενα επιτόκια ε, προφανώς ε, θα είναι και μεγαλύτερος κίνδυνος για να προκληθούν επιφυλάξεις και προβλήματα σχετικά με τη βιωσιμότητα. Θέλω να σας πω ότι όσον μέχρι πρόσφατα υπήρχε πρόβλημα σχετικά με τις μη μοχλευμένες δραστηριότητες και έχουμε διαπιστώσει ότι το 60% αυτών των ε, δανείων ε, κατέληγαν σε αθέτηση. Μιλάμε για ένα έξι φορές ε, μεγαλύτερο ποσό, πάνω από το έπιντα, κάτι που θα μπορούσαμε να δεχτούμε ως αποδεκτό επίπεδο. Ε, το Εποπτικό Συμβούλιο τον Μάιο του 2017 ήδη δημοσίευσε κάποιες ε, οδηγίες συγκεκριμένα να διευκολυνθεί ο εντοπισμός των μοχλευμένων συναλλαγών και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από έναν αρμονισμένο ή κοινό ορισμό έτσι ώστε τα στελέχη των τραπεζών να έχουν μία συνοπτική εικόνα ε, και να μπορούν να ε, προχωρούν και σε στοχευμένο έλεγχο. Ε, άλλα δάνεια που περνάνε έξι φορές πάνω από το έπιτα, αυτό θα πρέπει να είναι εξαίρεση ε, και θα πρέπει πάση θυσία να ε, παραπέμπονται σε μια ειδική επιτροπή. Αυτές, η εφαρμογή αυτών των οδηγιών της ε, ΕΚΤ έχουν άμεση σχέση με τα επίπεδα του GST, που έχει καθορίσει το GST, που εμείς τους ζητήσαμε να εξετάσουν αυτό το επίπεδο, έχουμε ξεκινήσει και συγκεκριμένες αποστολές για να ελεγχθεί το θέμα αυτό. Ως πρώτο αποτέλεσμα διαπιστώσαμε ότι ενδεχομένως να υπάρχει ε, μη ικανοποιητική εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών μας και ως εκ τούτου ε, θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε, ε, κατά πόσον η αντίδρασή μας θα πρέπει να είναι περισσότερο οριζόντια ή κατά πόσον θα πρέπει να εστιάζεται σε συγκεκριμένες τραπεζικές ενέργειες. Εν πάση περιπτώσει θα παρακολουθήσουμε το θέμα αυτό και επειδή είναι ένα θέμα ε, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας έχουμε έρθει σε επαφή με τους συναδέλφους μας που ασχολούνται με τη μακροπροληπτική ικανότητα για να έχουμε μια κοινή προσέγγιση ε, γιατί στο θέμα αυτό και η μακροπροληπτική ικανότητα θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό σημαντικό ρόλο. Όσον αφορά ε, την Συμφωνία Βασιλείας ε, και το πακέτο αυτό, νομίζω ότι ήδη ο πρόεδρος μας απάντησε σήμερα το πρωί λέγοντας ότι μαζί με την Κομισιόν θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας ε, στην οποία συμμετείχαμε και εμείς σε επίπεδο διαπραγματεύσεων. Και πιστεύουμε ότι η εφαρμογή σε μεγάλο βαθμό θα είναι ένα θετικό αποτέλεσμα. Όμως παρόλα αυτά ήδη υπάρχουν κάποιες αποκλήσεις. Ε, εμείς πιστεύουμε ότι οι αποκλήσεις δεν θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλες, αλλά στην εποπτική μας λειτουργία και δραστηριότητα θα λαμβάνουμε πάντα υπόψη μας την αναλογικότητα, όχι μόνο ε, το μέγεθος των τραπεζών, αλλά και το επιχειρηματικό τους υπόδειγμα. Ευχαριστώ πολύ. Λέει κύριος Φερνάντες. Θα μιλήσω ισπανικά. Τα τελευταία χρόνια ήδη μιλήσαμε πολύ για την ανάγκη βελτίωσης της Έλεγα λοιπόν ότι και στην Επιτροπή μας εδώ, αλλά και σε διάφορα φόρουμ ε, οικονομικής εποπτείας, συζητήθηκε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια η δυνατότητα να βελτιώσουμε την ε, εναρμόνιση όσον αφορά την τραπεζική αφαιρεγγιότητα, ώστε να έχουμε καλύτερες λύσεις. Και η συζήτηση αυτή για το μέλλον της εναρμόνισης στο θέμα ε, της αφαιρεγγιότητας οδήγησε και στη συζήτηση για ένα περισσότερο ασφαλές μέλλον ε, για τις αποτεμιεύσεις, το ευρωπαϊκό δηλαδή πρόγραμμα για την εγγύηση καταθέσεων. Και θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο που έχει να κάνει με αυτά τα δύο. Αλλά ίσως δεν ήταν πολύ συγκεκριμένη στην δημόσια συζήτηση. Πρόκειται για τις δυσκολίες ή για τις ρυθμίσεις που γίνονται για περιπτώσεις IPS ορισμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα συστήματα δηλαδή θεσμικής προστασίας κάποιων τραπεζών, είτε πρόκειται για από τα μιευτήρια που έχουν ορισμένες χώρες. Και οι παρεμβάσεις τους μπορεί να βοηθηθεί από εναλλακτικά μέτρα είναι αλήθεια όμως ότι τέτοιες παρεμβάσεις συχνά δεν ξέρουμε σε τι βαθμό μπορούν να θεωρηθούν κρατική ενίσχυση ή όχι. Έχουν γίνει διώξεις, έχουμε δίκες, αλλά η δυνατότητά τους να ε, μπορέσουν γρήγορα να έχουν κάποια βοήθεια από το κράτος, ενώ τα εθνικά συστήματα ασφάλειας καταθέσεων υφίστανται κάποια στρέβλωση. Όπως γίνεται και με τις ε, εθνικές ρυθμίσεις για την αφαιρεγκιότητα. Λίγο έχουμε συζητήσει για αυτά τα θέματα, παρόλο που θα ήταν σημαντικό να τα συζητήσουμε περισσότερο, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε καλύτερα στο μέλλον. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ για αυτήν την ερώτηση που και μας μας ενδιαφέρει πολύ. Γιατί ξέρουμε τι δυσκολίες αντιμετωπίζουμε εξαιτία των τεραστίων διαφορών που υπάρχουν ε, στις διάφορες χώρες όσον αφορά την αφαιρεγγιότητα των ε, τραπεζών. Ακόμα και λιγότερο σημαντικές ε, τράπεζες που θα λέγαμε ότι δεν εμποδίζεται η διάλυσή τους λόγω δημοσίου συμφέροντος. Αλλά ακόμα και εκεί έχουμε διαπιστώσει συχνά όταν έρθει η στιγμή πως τίθεται το θέμα της κρατικής ενίσχυσης. Γιατί σε κάποιες χώρες, σε περίπτωση ρευστοποίησης, μπορεί να υπάρχει βοήθεια, σε άλλες χώρες όχι. Τώρα, πέρα και από την σχετική οδηγία που λέει ότι υπάρχει υπάρχει ρευστοποίηση και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει κρατική βοήθεια, για μας αυτό είναι θετικό. Τώρα για τις παρεμβάσεις των IPS, αυτό είναι κάτι που συζητήθηκε πολύ στην περίπτωση Καρκάς, όπου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν επρόκειτο για κρατική ενίσχυση, ότι έγινε προς το συμφέρον ε, της τράπεζας, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε τα δικά της κριτήρια. Εξού και έκανε και έφεση. Τώρα θα πρέπει να παρακολουθήσουμε πάρα πολύ προσεκτικά γιατί υπάρχουν διάφορες δικαστικές υποθέσεις ε, με τις οποίες εξετάζεται η νομιμότητα ουσιαστικά. Γι' αυτό θα έλεγα ότι πράγματι υπάρχουν ε, θέματα με την παρέμβαση των IPS. Πρέπει να κάνει κάποιος μια διάκριση κατά πόσον υποχρεωτικά παρεμβαίνουν γιατί υποχρώνονται από τις κρατικές αρχές ή αν πρόκειται για παρέμβαση σε θελοντική βάση. Αλλά και πάλι θα έλεγα ότι όταν έχουμε την τελική απόφαση την οριστική του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα ξέρουμε περισσότερα. Μόνικα Σαμέντο, εκ μέρους του Renew. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω την ερώτησή μου στα γερμανικά, λουξεμβουργιέζικα δεν τα καταφέρνω. Αξιότιμη κύριε Μέσ, στην ομιλία σας πριν από δύο ημέρες μιλήσατε για την αποδοχή του Λίμπρα που από τις αρχές του 2020 προβλέπεται από το Facebook ως κυβερνονόμισμα. Αυτό το κυβερνονόμισμα, κατά τη γνώμη σας και κατά τη γνώμη της ΕΚΤ, αποτελεί κίνδυνο για την Ευρωζώνη γιατί θα, χάνει το, θα χάσει το μονοπόλιο του νομίσματος ε, η ΕΚΤ και θα έχει ε, ε, υψηλή σημασία και υψηλές επιπτώσεις για τις δραστηριότητε της ΕΚΤ και το ρόλο του ευρώ. το Φεβρουάριο του 2019 το Λουξεμβούργο, που είναι η χώρα προέλευσή σας, θέσπισε ένα νόμο για το blockchain, για την πρόθεση του blockchain. Οι πέντε γερμανόφωνοι υπουργοί συναντήθηκαν μεταξύ αυτών Γερμανία, Αυστρία, Λίχτενστάιν ε, και Λουξεμβούργο και σε αυτές τις νέες τεχνολογίες ε, συναλλαγών βλέπουν και κάποιες ε, ευκαιρίες αλλά και κάποιες προκλήσεις. Το Λίμπρα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκλεί τις συναλλαγές με το Λίμπρα και ξέρουμε ότι η Κίνα και άλλες δικαιοδοσίες επιτρέπουν το Λίμπρα. Αυτό θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να οδηγήσει σε κάποιο μειονέκτημα ανταγωνιστικό. Και ποιες είναι οι συνέπειες για την ε, Ευρωζώνη. Πώς θα πρέπει να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε αυτό. Και θα θέλετε μια ευρωπαϊκή λύση ή μια διεθνή λύση, παραδείγματο χάρη στα πλαίσια του ΟΣΑ για το Λίμπρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Η ομιλία μου πριν από δύο μέρες αφορούσε κυρίως ε, το χρήμα και τα trust. Μάλλον διορθώνω το χρήμα και την εμπιστοσύνη, γιατί είπα ότι ε, το χρήμα ε, έχει νόημα όταν το κοινό έχει εμπιστοσύνη στο νόμισμα που χρησιμοποιεί. Και γι' αυτό οι δημόσιοι οργανισμοί δεσμεύονται υπέρ του δημοσίου ωφέλους και τα ιδιωτικά νομίσματα που στοχεύουν στη μεγιστοποίηση των κερδών ε, μέσω της έκδοσης από ιδιώτες εκδότες δεν θα επιτύχουν το ίδιο επίπεδο εμπιστοσύνης όπως τα δημόσια νομίσματα. το Λίμπρα μπορεί να τεθεί ως νόμισμα το οποίο εκτοπίζει εθνικά νομίσματα, δημόσια νομίσματα. Υπάρχουν και άλλα θέματα σχετικά με την ε, ε, ε, ωφέλεια από πλευράς αποτελεσματικότητας και όταν υπάρχουν ωφέλη αποτελεσματικότητας τα χαιρετίζουμε ακόμη και όταν έρχονται από ιδιωτικές εταιρείες οι προσπάθειες αυτές που δεν προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. και ως εναλλακτική λύση θα μπορούσε να υπάρχει και κάποια ευρωπαϊκή λύση συγκρίσιμης αποτελεσματικότητας και ταχύτητας και που θα μπορούσαν να εκδίδονται από κεντρικές τράπεζες που έχουν δεσμευθεί υπέρ του κοινού ωφέλους. Σε μια σωστά λειτουργούσα οικονομία της αγοράς, η καινοτομία και οι καινοτόμες τεχνολογίες έχουν ως στόχο την πρόθεση όλων των φορέων τη οικονομίας της αγοράς που λειτουργεί σωστά. Από αυτή την οπτική γωνία λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ του Libra ως σταθερού νομίσματος και των κρυπτονομισμάτων. Το μόνο το οποίο μπορούν να έχουν ως κοινό γνώρισμα είναι ότι συχνά βασίζονται σε μια τεχνολογική πλατφόρμα που εμπνέεται από την τεχνολογία του blockchain. Κατά τα άλλα υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ ενός σταθερού νομίσματος και ενός κρυπτονομίσματος παραμένω σε αυτά τα οποία είπαμε, δηλαδή χαιρετίζουμε την καινοτομία και μέσα στις κεντρικές τράπεζες επίσης πειραματιζόμαστε με την καινοτομία και ενθαρρύνουμε τις ευρωπαϊκές λύσεις στον τομέα των πληρωμών, όπου προς το παρόν η Ευρώπη βασίζεται μόνο σε τεχνολογία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μεγάλο βαθμό. Τέλος, πιστεύουμε ότι οι κεντρικές τράπεζες είναι οι καλύτερα ενδεδειγμένες να εκδίδουν νομίσματα τα οποία θα χαίρουν τις εμπιστοσύνη του κοινού γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ. Ας έχουμε κατά νου το χρόνο για να μην παρατείνουμε τη διάρκεια της συνάντησης. Ο κ. Ρουτασάν, εκ μέρους των Πρασίνων. Κύριε Μέρς, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Καλησπέρα σας. Σε μία ομιλία στη Φραγκφούρτη τον Νοέμβριο του 2018 είχατε πει ότι η ΕΚΤ στενόμυαλα περιορίζει τις δυνατότητές της για να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή. Θεωρείτε ότι στο πρόγραμμα αγοράς ενεργητικού της ΕΚΤ και στο πρόγραμμα το εποπτικό θα έπρεπε να ασχοληθεί και με τη Συμφωνία του Παρισιού η ΕΚΤ και είχατε ε, τονίσει το πρόγραμμα αγοράς ε, στοιχείων ενεργητικού. Ε, αντίθετα με αυτό το οποίο μας είπε σήμερα το πρωί η κυρία Λαγκάρντ. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω στο ρόλο σας ως μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου, ως αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, βλέπετε την έκτη να μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο και τι δεσμεύσεις θα μπορούσατε να αναλάβετε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να διευκρινίσω ε, αυτό το θέμα, γιατί ποτέ δεν ήμουν υπέρμαχος της ε, χρήσης ε, στοιχείων ενεργητικού που έχουν σχέση με, το διοξίδι, με τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ως αντικείμενό της την προώθηση της σταθερότητας των τιμών και μπορεί να προωθεί αυτά τα οποία είναι περισσότερο αποτελεσματικά για το θέμα του κλίματος, αυτό το οποίο εννοούσα είναι ότι δεν έχουμε ηγετικό ρόλο στον προσδιορισμό μιας ταξινομίας, γιατί αυτό είναι αντικείμενο των νομοθετών. Αλλά από τη στιγμή που θα έχει οριστεί μια ταξινομία, για μας πολίτες της Ευρώπης, θα πρέπει εναπόκειται να υλοποιήσουμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρεπιπτόντως, συνεχίζουμε να επιθυμούμε να επικεντρωθούμε περισσότερο στην υλοποίηση. Αλλά δεν μπορούμε να τα προσδιορίσουμε εμείς. Αυτό είναι πέραν της δικής μας εντολής. Αυτό ήταν το αντικείμενο της ομιλίας μου τότε. Επίσης, θα θέλαμε να έχουμε καλύτερες κατευθυντήριες γραμμές από τις αρμόδιες αρχές για τη διάκριση μεταξύ πράσινων στοιχείων ενεργητικού και βιώσιμων στοιχείων ενεργητικού. Γιατί μερικές φορές για μας είναι δύσκολο να κατανοήσουμε αν μια επένδυση σε πυρηνική ενέργεια θεωρείται πράσινη ή θεωρείται και βιώσιμη δεν είναι ρόλο τη ΕΚΤ, ούτε στη λειτουργία της για την νομισματική πολιτική, ούτε στη λειτουργία της για την εποπτεία, να υποκαταστήσει τι αρμοδιότητες του νομοθέτη. Σα ευχαριστώ πολύ. Γκούναρ Μπέκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Μέρσο. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ε, η κυρία Λαγκάρτ που ίσως ε, ε, θα είναι και ε, προϊσταμένη σας, ήταν σήμερα εδώ το πρωί. Η κυρία Λαγκάρτ μέχρι τώρα είναι η μόνη πολιτικός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα σε διεθνές επίπεδο που δέχεται ότι η ΕΚΤ και άλλοι παραβίασαν τους, τις συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης για να σώσουν το ευρώ. τώρα, η κυρία Λαγκάρτ για το μέλλον είπε ότι το να υπάρξουν άλλες ε, παραβιάσεις, transgressions μίλησε κατά λέξη, αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε, τέτοιου είδους ε, παραβιάσεις ε, ε, δεν θα πρέπει να λάβουν χώρα. Αν ε, είχατε γενέθλια ή αν είχαμε Χριστούγεννα, ε, τι θα ευχόσασταν σχετικά με αυτό το ενδεχόμενο, το να μην υπάρξουν άλλες παραβιάσεις προς όφελος του κοινού συμφέροντος για τα επόμενα πέντε χρόνια. Thank you for the question. I have heard uh, Σας ευχαριστώ πολύ. την παρακολούθησα την ακρόση με την κυρία Λαγκάρτ και πρέπει να ομολογήσω ότι δεσμευόμαστε από το κράτος δικαίου και ο έλεγχος των ευρωπαϊκών θεσμών. Ε, δεσμευόμεθα επίσης από τους θεσμούς που ορμηνεύουν το δίκαιο, δηλαδή από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ορισμένες από τις ε, αποφάσεις μας ε, υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει επιβεβαιώσει συγκεκριμένες αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Η δεύτερη ήταν η περίπτωση Vice. Και στις δύο περιπτώσεις ε, ο φυσικός μας δικαστής, το κανονικό δικαστήριο, αποφάσισε ότι δεν παραβιάσαμε τα όρια της εντολής μας. Δεν προχωρήσαμε πέρα από αυτά, αλλά παραμείναμε μέσα σε αυτά τα όρια της εντολής και διότι το ε, δικαστήριο αναγνώρισε ότι Υπάρχουν ε, κάποιοι περιορισμοί και το δικαστήριο είπε ότι λειτουργήσαμε με σωστό τρόπο, αναλογικό και επίσης ε, κάναμε μια ικανοποιητική ανάλυση κόστους-οφέλους για να διαπιστώσουμε κατά πόσον ε, οι επιθύμητες αρνητικές συνέπειες θα μπορούσαν να αντισταθμιστούν από θετικές ε, ναι, προεκτάσεις. Ως εκ τούτου, ε, εμείς θεωρώ ότι καλύπτουμε τις προϋποθέσεις που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και δεν νομίζω ότι καμία στιγμή ξεφύγαμε από την εντολή μας, γιατί ξέρετε εμείς αυτό δεν το συνηθίζουμε. Πολύ ωραία. Επόμενος Μιλητή ε, ρωτών από το ECR. Ευχαριστώ πολύ. Στα Ολλανδικά θα υποβάλω την ερώτησή μου. Έχετε εμπειρία από τις τράπεζες, ε, ήδη το 2012 ήσασταν στο Εράσμος και θέλω να σας ρωτήσω εσείς τώρα πώς βλέπετε τις εξελίξεις ε, μετά την κρίση της Ευρωζώνης την οποία ζήσατε κι εσείς. Η κρίση στο ευρωσύστημα ήταν βαθιά. Εσείς θα είχατε κάνει κάτι διαφορετικά. Τι διαφορετικό θα είχατε κάνει. Και η Ευρωζώνη με τις ε, εξελίξεις στη νομισματική ένωση είναι αυτή που θα μας οδηγήσει στην επόμενη κρίση. Ουσιαστικά πρόκειται για τον προβληματισμό. Πώς δηλαδή ε, αξιολογείτε εσεί τα χρόνια που πέρασαν και τι μαθήματα πήρατε από την εμπειρία των τελευταίων ετών για να ασκήσετε τα καθήκοντά σας στο μέλλον. Επιτρέψτε μου να απαντήσω πρώτα τη δεύτερη ερώτηση. Γιατί πάντα στην ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, λέμε ότι η απόφαση είναι αυτών που χρησιμοποιούν την υπηρεσία μας και όταν υπάρχει κάποιο αίτημα για κάποια άδεια εμείς συνεχίζουμε να προσφέρουμε ασφαλή εργαλεία. Αν βέβαια υπήρξε αυξανόμενη ζήτηση για άλλου είδους τεχνολογική στήριξη για να χρησιμοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τότε θα μπορούσαμε να είμαστε έτοιμοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα για τέτοιο διαφοροποιημένο μέσο. Πάντα προσπαθούσαμε να είμαστε ιδιαίτερα αποτελεσματικοί προκειμένου να ικανοποιούμε τα αιτήματα των πολιτών όταν πρόκειται για τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για το πρώτο τώρα ερώτημα. Η Ευρωζώνη σε πολιτικό επίπεδο έχει δείξει ιδιαίτερα η υψηλό επίπεδο δέσμευσης να κρατήσει το ευρώ, αυτό το λέω βλέποντας τα πράγματα από μέσα, ε, πολύ περισσότερο από ότι αν κάποιος θα βλέπει τα πράγματα απ' έξω. Τώρα, αν θα είχαμε τα νιώσει για κάτι, ίσως ότι δεν κάναμε περισσότερα και πιο γρήγορα. Και αν είχαμε ολοκληρώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήταν καλύτερα Παρόλα αυτά, σε κάθε περίπτωση θα μένανε κάποια στοιχεία της ε, Τραπεζικής Ένωσης χωρίς να είναι ολοκληρωμένα, αλλά αυτό που θα έπρεπε να έχουμε κοιτάξει περισσότερο και να το κάνουμε και τώρα είναι η αρχιτεκτονική της Τραπεζικής Ένωσης. Οι συζητήσεις πάντως έχουν προχωρήσει πολύ και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Όμως πρέπει ακόμα να ξεπεράσουμε την διάκριση αυτή του επιμερισμού κινδύνου και της μείωσης του κινδύνου. Στο θέμα της τραπεζικής εποπτείας, όταν μιλάμε για την μείωση του κινδύνου, το είπα και στην αρχή και το είπε και ο πρόεδρος Ενρία σήμερα το πρωί, έχει επιτευχθεί τεράστια πρόοδος. Έχει μειωθεί ο κίνδυνος και έχουμε ετοιμάσει και το πλαίσιο για να ελέγχουμε μελλοντικού κινδύνους. Οπότε τι μαθήματα έχουμε πάρει. Πίστευω ότι τώρα είμαστε έτοιμοι να μπορέσουμε να δράσουμε πιο γρήγορα. Ολοκληρώνοντας την Τραπεζική Ένωση, για παράδειγμα το σκέλος για την εγγύηση καταθάσεων. Συγχρόνως και για την ρύθμιση όσον αφορά την ε, έκθεση σε ομόλογα, σε κρατικά ομόλογα. Σίγουρα χρειάζεται συζήτηση και για το μέγεθος του ενεργητικού. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία εκδίδει η ίδια στοιχεία, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να συζητηθεί περισσότερο. Πάντως υπάρχουν διάφορα ρεύματα συζήτηση και θα έπρεπε εκ παραλίλου να γίνονται οι συζητήσεις αυτές, ώστε η αρχιτεκτονική μας να είναι πιο ε, αποτελεσματική. Αυτό θα ήταν βέβαια ευπρόσδεκτο εν ώψη οποιασδήποτε νέας κρίσης. Τώρα, από την ΚΟΕ, δεν ξέρω, θέλει κάποιο να λάβει το λόγο από την ΚΟΕ. Αν όχι, ε, τότε για τον επόμενο γύρο ε, θα έχουμε πρώτα την κυρία Ντανούτα Χούπνερ από το ΕΛΚ. Κοιτάξτε, ε, το πρόβλημα μου είναι ότι μόλις τώρα απαντήσατε στο ερώτημα που ήθελα να σας δέξω. Γιατί εγώ ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τη ρυθμιστική αντιμετώπιση του κρατικού χρέους. Να το πω αλλιώς. Συμφωνείτε μαζί μου ως προς το ότι θεωρητικά υπάρχουν ε, θετικές επιπτώσεις ε, όσον αφορά ε, τα κεφάλαια αυτά στον, προ, στην πρόοδο προς την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Η εξασφάλιση των καταθέσεων ε, πράγματι είναι μια δυνατότητα και για να μειωθεί το κρατικό χρέος, εγώ πιστεύω ότι αυτά τα κεφάλαια θα μπορούσαν να μειώσουν κάπως τους κινδύνους. Αλλά κατά την άποψή σας, ποιες είναι οι δυνατότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Ε, αυτή είναι μια ερώτηση και ίσως μπορείτε και να ε, σχολιάσετε σε αυτά που είπατε. Ε, το δεύτερο ερώτημά μου είναι το εξής. Ας ελπίσουμε ότι τα επόμενα έτη ε, δεν θα έχουμε ύφεση στην Ευρώπη, θα έχουμε απλά μια επιβράδυνση, ε, πιο δύσκολη οικονομική κατάσταση και για πρώτη φορά ε, τόσο ο εποπτικός μηχανισμός όσο και ο μηχανισμός εξυγίανσης θα λειτουργήσουν την εποχή, τη στιγμή που θα έχουμε ύφεση. Εσείς πώς ακριβώς αξιολογείτε την αντίσταση, την ανθεκτικότητα των οργανισμών που φτιάξαμε ε, στην Ευρώπη μετά την κρίση. Αυτοί οι μηχανισμοί θα μπορούσαν να βοηθήσουν έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί καλύτερη κρίση από ό,τι συνέβη μέχρι σήμερα. Εγώ ε, δεν ε, αμφισβητώ επουδενή την καλή βούληση, την θέληση και την ενέργεια που εκφράστηκαν από πολλούς. Υπάρχει βέβαια και το στοιχείο της εμπιστοσύνης. Για κάποιους ανθρώπους εμπιστοσύνη οικοδομείται σιγά σιγά, γι' αυτό και αυτές οι συζητήσεις ε, ε πολλές φορές ε, παρατείνονται. Βέβαια δεν μπορούν να παρατείνονται στο διηνεκές μέχρι να έρθει και η επόμενη κρίση. Σήμερα το πρωί η υποψήφια για την Προεδρία της ΕΚΤ είπε ότι έχει ε, διαπιστώσει ότι η Ευρώπη είναι στα καλύτερά της όταν είναι στα χειρότερά της. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι σε περίοδους κρίσης σημειώνουμε ουσιαστική πρόοδο. Και είπε επίσης ότι ελπίζει εκείνη να προσφέρει μια εναλλακτική λύση σε αυτή την ε, πρόοδο και συμφωνώ μαζί της. Ειλικρινά πιστεύω ότι το θεσμικό πλαίσιο ε, που προτείναμε, το θεσμικό αυτό πλαίσιο βοηθάει στην ανθεκτικότητα ε, στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη. Και αυτό έχει πολλές ε, διαστάσεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε ικανοποιημένοι και ότι πρέπει και μπορούμε να προσφέρουμε εγγύηση ότι όταν θα χτυπήσει η κρίση θα είμαστε έτοιμοι. Τώρα όμως ε, έχουμε τουλάχιστον έτοιμους τους θεσμούς. Κατά τη διάρκεια της ε, τελευταίας κρίσης ε, είχαμε φτιάξει το σπίτι, αλλά δεν είχαμε ε, πυροσβεστικές δυνάμεις για περίπτωση ανάγκης. Τώρα έχουμε πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά δεν ξέρουμε αν αρκούν αυτές. Ε, υπάρχει βέβαια εμπειρία από την προηγούμενη κρίση. Αυτό είναι κάτι θετικό. Ένα κομμάτι της ερώτησης ε, αφορά στο τι λείπει ακόμα. Αυτό που δεν έχουμε ακόμα πλήρως ε, είναι δεν έχουμε ρυθμίσει το θέμα της ρευστότητας και της εξυγίανσης και ποιος θα είναι αρμόδιος για αυτά τα δύο. Αν δούμε το τι συμβαίνει, παραδείγματο χάνει στι Ηνωμένε Πολιτείε, εκεί υπάρχει ε, το FDIC, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι το FDIC, όπως συμβαίνει και με την Τράπεζα της Αγγλίας, έχει απόλυτη απόλυτες εγγυήσεις για, για ρευστότητα και εξυγίανση αυτό το εγγυάται το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ. Στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε κεντρικό Υπουργείο Οικονομικών, άρα πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις. Θα πρέπει, παραδείγματος χάρη, να δώσουμε ε, στις ε, ε, συστημικές τράπεζες ή στις κεντρικές μάλλον τράπεζες ε, μεγαλύτερη πρόσβαση στα χρήματα της ΕΚΤ από ό,τι έχουν οι απλές τράπεζες. Επαρκή εχέγγυα. Άρα κατά άποψή μας η εγγύηση που θεωρούμε ότι είναι επαρκής ε, θα πρέπει να είναι η ικανοποιητική κάλυψη τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων, γιατί ε, μόνο έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη ρευστότητα. Καλύτερα να σταματήσω εδώ και να μην μπω σε περισσότερες ε, λεπτομέρειες. Έχω άλλη μια ερώτηση για τους σοσιαλδημοκράτες. Δεν βλέπω κάποιον. Ο Γιώνας ε, θέλει να κάνει μια ερώτηση. Πάνω από ένα χρόνο τώρα είχαμε το θέμα της Ισπανικής Τράπεζας Banco Popular. Και ακόμα και χτες διαβάζαμε ότι οι προηγούμενες αναλύσεις όταν είχε υπάρξει ενημέρωση ξέραμε ότι υπήρχαν στα Μητρό οι αναλύσεις οι Σήμερα διαβάσαμε σε κάποια μέσα ενημέρωσης ότι σε περίπτωση ε, στρες τελικά είχαν υποτιμηθεί η δυνατότητα διατήρησης ρευστότητας ε, κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Το θέμα αυτό της ρευστότητας είναι που οδηγεί σε αφαιρεγκιότητα όπως έγινε και σε αυτή την περίπτωση. Κατά τη γνώμη μου όμως, όταν υπάρχει μια κρίση ρευστότητας, προηγείται μια κρίση σαφερεγκιότητας, που είναι κάπως και καλυμμένη. Οπότε, ενώ οι κρίσεις ρευστότητα οδηγούν σε ενώ για μένα πρώτα έρχεται η αφαγγερότητα και μετά η κρίση ρευστότητα. Από αυτά που γνωρίζουμε σήμερα και από τις προηγούμενες αναλύσεις που έχουμε σε περίπτωση δοκιμών ε, αντοχής, στη θεωρία θα έπρεπε να είχε παραπάνω περίπου 2 δισεκατομμύρια για να αποφύγει την κρίση η τράπεζα. Έγιναν δηλαδή λάθη εποπτείας και αποφάσιστηκε η εξυγένση μέσα σε λίγες ώρες, αλλά υπήρχαν προβλήματα εποπτείας, τα οποία επέτρεψαν στην τράπεζα αυτή να παραμένει με προβλήματα αφαιρεγγιότητας και καλυμμένο, όπως είπα και πριν. Είναι λοιπόν σημαντικό να αναθορίσουμε, να ξαναδούμε λίγο πώς γίνονται αυτές οι δοκιμές ε, αντοχής και σχέση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών με τον SSM για να μην ε, κρύβονται προβλήματα όπως πιστεύω ότι έγινε στην περίπτωση της ΠΑΝΚΟ Ποπουλάρ, που πιστεύω ότι θα μπορούσε να είχαν πολύ πιο εύκολα. Το πρόβλημα ήταν ότι υπήρχε και καλυμμένη αφαιρεγκαιότητα στην περίπτωση αυτής της τράπεζας πριν εμφανιστεί το πρόβλημα της ρευστότητα. Ευχαριστώ. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να σχολιάσω με λεπτομέρειες την περίπτωση αυτή. Τότε Ήμουν μόνο στην νομισματική πτυχή. Και αυτό το οποίο είναι γνωστό, ότι το ότι πήγαινε για χρεοκοπία ή σχεδόν για χρεοκοπία, οφείλεται στην έλλειψη ρευστότητας και όχι σε αφαιρεγγιότητα. Η τράπεζα τότε οχι σε αφαιρεγκαιοτητα η όλες τις ε, μακροπροληπτικές ε, προϋποθέσεις, δηλαδή είχε το κεφάλαιο που χρειαζόταν και ανταποκρινόταν στον ορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων σύμφωνα με την εποπτική αρχή και με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Τώρα, ε, το, η δοκιμή αντοχής δεν ήταν το μόνο στοιχείο. Ήταν και το διαθέσιμο κεφάλαιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχε ο επόπτης. Η τράπεζα φαίνεται να ανταποκρινόταν στις προϋποθέσεις έτσι όπως είχαν καθοριστεί νωρίτερα. Τώρα, η δοκιμή αντοχής έγινε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Και το SSM, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, Κεντρική Τράπεζα, μόνο μακροοικονομικά σενάρια παρουσιάζει. Από αυτή την άποψη λοιπόν δεν είναι αυτό ένα στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να είχε εντοπίσει την αφαιρεγκιότητα παρόλο που είναι αλήθεια ότι ήδη τότε η εν λόγω τράπεζα δεν ήταν από αυτές που είχε τις καλύτερες επιδόσεις. Ήταν μάλλον σε χαμηλό επίπεδο επιδόσεων μετά τις δοκιμές αυτές αντοχής. Αλλά ήταν πάνω από το όριο πάντως. Οπότε, από όσο γνωρίζω εγώ και γνωρίζω αυτά τα οποία είναι δημόσια, δεν υπήρχε καμία ένδειξη η οποία να μας οδηγούσε ε, στο συμπέρασμα για αφαιρεγκαιότητα και ήταν η κρίση ρευστότητα η οποία μας έκανε να κρίνουμε ότι η τράπεζα αυτή πήγαινε για χρεοκοπία ή σχεδόν χρεοκοπία. Και πάλι ζητώ συγγνώμη επειδή μιλώ βάσει των όσων γνωρίζω και τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε. Ωραία. Ε, ολοκληρώνουμε εδώ. Είμαστε στην ώρα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε ε, σήμερα και απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις μας. Ευχαριστώ όλους και για την ε, πειθαρχία. Ένα λεπτό θα διακόψουμε για να συνεχίσουμε με το επόμενο θέμα και με τον συνάδελφο Μουρισάν. Can I ask you to get back to your seat so that we can start? Είστε παρακαλώ για να μπορέσουμε να αρχίσουμε. Κοντεύουμε, κοντεύουμε. Λοιπόν, συνάδελφοι, ε, όσοι θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση θα πρέπει να έχουν έρθει ήδη. Ε, πρόκειται για το Γενικό Προπλογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Οικονομικό έτος 2020, όλα τα τμήματα. Ε, ε, και συντάκτης είναι ο Σίκφριτ Μούρεσαν και τώρα ε, νομίζω θα εξετάσουμε κάποιες τροπολογίες. Δεν ξέρω τι θα πρέπει να πω, αλλά η πρακτική είναι να έχουμε την άποψη της ΕΚΟΝ και από την άλλη της ε, τροπολογίες. 25 Ιουλίου ήταν η ημερομηνία κατάθεσης ε, τροπολογιών. Ε, θα πρέπει να υπάρχουν ικανοποιητικοί πόροι για μακροοικονομικές πολιτικές, όπως επίσης και ικανοποιητικοί πόροι για τις ίδιες τις ευρωπαϊκές αρχές. Η ανταλλαγή απόψεων είναι η εξή. Ο εισηγητή έχει τρία λεπτά για να παρουσιάσει την πρότασή του και μετά οι σκιώδεις εισηγητέ ε, δύο λεπτά και αν χρειαστεί θα πάμε στο Catch the Eye. Ε, καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι ε, και εγώ να σας ε, καλωσορίσω να σας εξηγήσω λίγο τι ακριβώς σημαίνει αυτή η γνωμοδότηση της ΕΚΟΝ για το 2020. Κάθε χρόνο την Άνοιξη κανονικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέτει το σχέδιο προεπολογισμού για την επόμενη χρονιά και το Συμβούλιο τοποθετείται από αυτού. Κανονικά το Συμβούλιο κάνει περικοπές στο σχέδιο προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά πρέπει να τοποθετηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και κάνουμε ε, έχουμε το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και μερικές φορές είμαστε παραπάνω, πιο πάνω, γιατί εμείς ως ε, Κοινοβούλιο λέμε το εξή. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί αποφασίζουν ποιε είναι οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητάμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει όλο και περισσότερα και αυτό το ζητάνε πολλές φορές και οι κυβερνήσεις. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται έναν προπολογισμό που να ε, καλύπτει τις αρμοδιότητες και γι' αυτό ε, Συνήθω εμεί προτείνουμε υψηλότερο προπολογισμό. Και επειδή πάντα είναι διαφορετική η θέση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γίνεται η τελική συνδιαλλαγή για να αποφασιστεί ο προπολογισμό. Είμαστε τώρα στην εξή φάση. Το Συμβούλιο έχει αποφασίσει για τη θέση του. Το Κοινοβούλιο καλείται τώρα να αποφασίσει για τη θέση του. Η Επιτροπή που λαμβάνει τι αποφάσει είναι η Επιτροπή Προπολογισμών και πριν αυτή η Επιτροπή αποφασίσει τέλη Σεπτεμβρίου, αρχέ Οκτωβρίου, όλε οι άλλε επιτροπέ ε, πρέπει να ε, καταθέσουν τις γνωμοδοτήσεις τους, ελπίζοντας ότι αυτές θα ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή Προεπολογισμών. Και εγώ ε, πρέπει να σας πω, όταν ήμουνα το 18 εισηγητή, ε, εξέτασα πολύ προσεκτικά αυτές τις γνωμοδοτήσεις και προσπάθησα να συμπεριλάβω όσο δυνατόν περισσότερα. Άρα δηλαδή η δουλειά μας ε, παίζει ρόλο τον Ιούλιο παρουσίασα τις τροπολογίες. Εσείς είχατε τη δυνατότητα επίσης να καταθέσετε. Τώρα συζητάμε για τις τροπολογίες και σήμερα το βράδυ θα εξεταστούν ε, οι τροπολογίες. Δεν θα μιλήσω πάλι για την έκθεση. Εγώ θα τοποθετηθώ μόνο επί των τροπολογιών που κατέθεσαν οι ε, συνάδελφοι. 38 κατατέθηκαν και 48 τροπολογίες στις γνωμοδοτήσεις. Ξεκινάω με τις ε, τροπολογίες του προϋπολογισμού, γιατί αυτές είναι και πιο σημαντικές. Το πλαίσιο ε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι οι οργανισμοί που εμπίπτουν στις δικές μας τις αρμοδιότητες. Η Κομισιόν έχει προτείνει ένα συγκεκριμένο ποσό, το Συμβούλιο προτείνει περικοπές, εγώ λέω το εξή. Θα ήθελα ως Κοινοβούλιο να απορρίψουμε τις ε, περικοπές του Συμβουλίου. Είμαι σε πολύ στενή επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης είμαι μέλος ε, του θεσμικού φορέα για τους εξωτερικούς αυτούς οργανισμούς και οι προτάσεις που κάνει η Κομισιόν στο σχέδιο του προπολογισμού είναι λογικές. Ούτε πολύ ψηλές, ούτε πολύ χαμηλές. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι πρέπει να απορρίψουμε τις περικοπές του Συμβουλίου, γιατί αυτό θα επηράσει τη δουλειά των εξωτερικών οργανισμών. Και όσοι συνάδελφοι λένε να αυξηθούν οι προπλογισμοί των εξωτερικών οργανισμών, τους λέω ε, μίλησα με τους οργανισμούς αυτούς, μίλησα με τις υπηρεσίες ε, της ε, ε, εποπτικής αρχής για τους φορείς, για τους εξωτερικούς οργανισμούς. Και αυτή τη στιγμή ε, θέλω να σας πω ότι ε, δεν ζητούνται αυξήσεις αυτών των οργανισμών, αλλά όχι αύξηση των κοντιλιών. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ προτείνω να ζητήσουμε για αυτούς τους ε, οργανισμούς και αυτές τις αρχές ε, τα, τα ποσά τα οποία προτείνουμε εμείς. Βεβαίω, ε, ξέρω τι συμβαίνει με τις εποπτικές αυτές αρχές. Και Πολύ συχνά λοιπόν ε, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτά είναι επιθυμίες αυτών των ε, οργανισμών, των φορέων και ε, δεν ξέρουμε κατά πόσον βασίζονται στις πραγματικές ανάγκες. Πάντως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τον προϋπολογισμό μας. Κλείνω αυτό το κεφάλαιο. Η δική μου πρόταση είναι να δεχτούμε την πρόταση της Κομισιόν σχετικά με αυτούς τους φορείς. Οι συνάδελφοι κατέθεσαν κάποιες ε, τροπολογίες για να ε, μπουν ε, κάποιες γραμμές σε απόθεμα. Εγώ συμφωνώ με αυτήν την προσέγγιση και γι' αυτό συμφωνώ με την προφορική τροπολογία του συναδέλφου Σβέν Γκίγκολτ, που είναι σε απόθεμα να μπουν οι γραμμές που αφορούν στον, στους ελέγχους ε, γιατί ε, ο πρώην συναδελφός μας, ο Τολοζάν, ήταν που κατάρτισε μία έκθεση μέσα από τις οποίες ζητάμε από τις αρμόδιες αρχές να εφαρμόζουν αυτά που ζητάμε όσον αφορά ε, τους ελέγχους, τους δημοσιονομικούς ελέγχους. Ε, τους λέμε τα χρήματα που σας δίνουμε θα πρέπει να τα βάλετε σε απόθεμα. Αυτή είναι η πρώτη τροπολογία και η δεύτερη τροπολογία που στηρίζω είναι ε, να βάλουμε κάποιες γραμμές της Eurostat σε απόθεμα. Εκτιμώ τη δουλειά της Eurostat αλλά οποτεδήποτε θέλω κάποιες ε, πληροφορίες για τη Eurostat. Ε, είναι πάρα πολύ περίπλοκη η διαδικασία. Η Eurostat λοιπόν πρέπει ε, τη δουλειά τους να την προσαρμόσουν περισσότερο στους χρήστες. Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε χρόνο είναι 74 εκατομμύρια ευρώ και οι τροπολογίες λένε 4 εκατομμύρια να πάνε στο απόθεμα. Πολύ είναι, εγώ λέω 2 εκατομμύρια ευρώ. Το πολιτικό μήνυμα όμως είναι ότι θα πρέπει να τους εξηγήσουμε ακριβώς ε, γιατί θα πρέπει να το κάνουν αυτό και γιατί πρέπει η δουλειά τους να είναι πιο φιλική προς τους ε, χρήστες, κυρίως και για το ευρύτερο κοινό. Τρίτον, υπάρχει πρόταση 90 εκατομμύρια ευρώ από τις ε, εγγύσεις, αυτά να πάνε σε απόθεμα. Αυτό αφορά ε, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Εδώ προτείνω να καταψηφίσουμε και θα σε εξηγήσω γιατί διαφωνώ. Το πρόγραμμα στρατηγικών επενδύσεων λειτουργεί, ε, οδηγεί σε περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες θέσεις απασχόληση στην Ευρώπη. Ε, δεν θα πρέπει να δώσουμε κάποιο αρνητικό μήνυμα στις αγορές. Γνωρίζουμε ότι το σύστημα δουλεύει, δεν είναι τέλειο, ίσως θα πρέπει να βελτιώσουμε τη σωρευτικότητα των προγραμμάτων. Εγώ από τη Ρουμανία θέλω να σας πω ότι οι εκλογής μου με ρωτάνε γιατί τόσες πολλές επενδύσεις πάνε σε άλλες αναπτυγμένες χώρες και σε εμά πολύ λιγότερο, γιατί έχουμε ε, μειονεκτήματα. Οι κεφαλοαγορές μας δεν είναι αναπτυγμένες. Η εμπειρία μας με τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία είναι περιορισμένη. Άρα δηλαδή το ΕΦΣΥ θα πρέπει να βελτιωθεί κυρίως όσον αφορά την τεχνική αρρωγή και την βοηθεία προς ε, νέες χώρες. Γίνονται όμως αυτά και γι' αυτό προτείνω ότι δεν χρειάζεται τώρα να αμφισβητήσουμε το ΕΦΣΥ βάζοντας ένα τόσο μεγάλο ποσό σε απόθεμα. Και τρίτον, και αυτό είναι το τελευταίο που θέλω να πω, αφορά σε πιλωτικά προγράμματα και ε, προπαρασκευαστικές ε, πράξεις. Ε, τον Ιούλιο είπα σε μία συνάντηση ότι όσον αφορά αυτές τις ε, πράξεις. Ε, έστειλε στην ε, Επιτροπή ένα εγγραφό για αξιολόγηση και η Επιτροπή θα αποφασίσει κατά πόσον χρειάζονται ίσως μικρές αλλαγές. Να δει επίσης η Επιτροπή κατά πόσον όλα αυτά ήδη καλύπτονται από άλλη δουλειά της Επιτροπής. Εγώ λοιπόν θα λάβω υπόψη μου μόνο ε, προγράμματα που βαθμολογούνται με α ή β και γι' αυτό το λόγο προτείνω να συστήριξουμε επιλογικά προγράμματα με βαθμολογία α ή β. Υπάρχει η πρόταση να ε, δημιουργηθούν νέες δομές ε, σχετικά με την καταπολέμηση του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Ε, υπάρχει ήδη ένα σχετικό πρόγραμμα όμως για αυτό το θέμα, το πρόγραμμα Φισκάλης. Και γι' αυτό πιστεύω ότι ένα επιπρόσθετο πιλωτικό πρόγραμμα δεν δικαιολογείται ε, το να εστιάζουμε σε πολλά διαφορετικά, δεν είναι σωστό, ας πάμε σε αυτό που έχουμε. Και υπάρχει και το πρόγραμμα εκείνο όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις ε, προκήρυξε διαγωνισμό για μελέτη για αυτό το θέμα. Άρα δηλαδή και αυτή η δουλειά καλύπτεται Αυτά είχα να σας πω για τις ε, τροπολογίες προϋπολογισμού και όσον αφορά το κείμενο της ε, γνωμοδότησης ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι ασχολήθηκαν με τη δουλειά αυτή. Έχουμε καταθέσει τέσσερις τροπολογίες για τα πιο σημαντικά θέματα για την ανταγωνιστικότητα των επενδύσεων ενώ διαφυλάσσεται το σύμφωνο σταθερότητας, καταπολέμηση του ξεπλήματος, φοροδιαφυγή και Τέλος, η ανάγκη να χρηματοδοτούμε σωστά τους ε, φορείς ε, ΕΖΑΣ. Ε, νομίζω συμφωνήσαμε όλοι για αυτούς τους τέσσερις συμβασμούς και θα ήθελα να συμφωνήσουμε όλοι. Αυτά είχα να σας πω και προσβλέπω στις συζητήσεις και στην ψηφορία που θα λάβει η χώρα σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ για την εισαγωγή αυτή, το τρίλεπτη, όπως προβλεπόταν, που έγινε ενδεκάλεπτη. Δεν θα προλάβουμε να ψηφίσουμε αργότερα, αν συνεχίσουμε έτσι. Δύο λεπτά, παρακαλώ. Γιώνας, ευχαριστώ πολύ. Θα είναι πολύ σύντομο. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, ο οποίος σε σύντομο χρονικό διάστημα πρότεινε συμβιβασμούς που ευχαρίστως να υπερψηφίσω εφόσον ληφθούν υπόψη τα σχόλια της ομάδας μου. Βλέπω ότι πολλές από τις τροπολογίες στηρίζουν κοινωνικές δράσεις. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο πράγματι θα πρέπει να αποτελεί ένα μέσο για την υλοποίηση του έντης. Τώρα για άλλες τροπολογίες. Εμείς στηρίζουμε τις τροπολογίες του εισηγητή για να επανέλθει το σχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τα μέσα να εργαστεί και να εποπτεύσει όλες τις μεταρρυθμίσεις. Μαζί με τους συναδέρφους προτείνουμε ένα νέο προπαρασκευαστικό παράρτημα το οποίο θα συνοδεύσει τα όσα έχει εφαρμόσει μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τάξη πρέπει να μπορέσει να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο και τίποτα άλλο. Θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον κύριο Μούρεσαν για την καλή συνεργασία που είχαμε τις τελευταίες εβδομάδες. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε Renew. Λουί Ριγκάνο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τον εισηγητή για το έργο του που καλύπτει τις κύριες ανησυχίες νομίζω της Επιτροπής μας. Ευχαριστούμε που λαμβάνετε υπόψη σας τα σχόλια της ομάδας μας και τα έχετε ενσωματώσει στις συμβαστικές τροπολογίες. Πιστεύουμε ότι ο προπολογισμός του 2020 πρέπει να περιλαμβάνει τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και να βοηθήσει τον συντονισμό, την εποπτεία και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε το οικονομικό έγκλημα επίσης. Τέλος, αντιλαμβάνομαι τις προκλήσεις των εποπτικών αρχών που δεν έχουν αρκετή πρικοδότηση είναι πολύ σημαντικές γιατί είναι αναγκαίες προκειμένου να υποπτεύουν την τήρηση των κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά την φορολόγηση, πρέπει να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή. Οπότε εννοείται ότι το στηρίζουμε όπως επίσης και το παρατηρητήριο. Εγώ και οι άλλοι συνάδελφοι από το Ρινιού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Σβέν Γκίγκολτ, μέρο των Πρασίνων. Ευχαριστώ. Ναι, και εγώ. Θερμές ευχαριστίες στον εισηγητή για την καλή συνεργασία που είχαμε μεταξύ μα και το ευρωπαϊκό πνεύμα που υπερίσχυσε προκειμένου να καταλήξουμε στις προτάσεις αυτές. Ε, περιγράφει η γνωμοδότηση πολύ καλά πώς λάβαμε υπόψη, πώς λήφθηκαν υπόψη οι δικές μας παρατηρήσει, οπότε το στηρίζουμε. Τώρα, πάντα οι φορείς θέλουν περισσότερα. Εδώ όμως υπάρχει μια διαφορά. Γιατί ολοκληρώθηκε η έκθεση με τον Ότμαντ Κάρας για την μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής. Με το ίδιο πνεύμα. Συνεπώς, Συμφωνώ με τους άλλους συναδέρφους ότι η αύξηση του προπολογισμού πρέπει να ακολουθήσει τα όσα αιτιολογεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει κάποιες αλλαγές, ε, γίνονται δεκτές, αλλά μετά δεν υπάρχει η αντίστοιχη πρικοδότηση. Οπότε γίνεται σκληρή δουλειά με ελάχιστο προσωπικό από τις υπηρεσίες αυτές. Αιτιολογείται να αυξηθεί ο προπολογισμό τους. Φυσικά μετά θα πρέπει να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο, εννοείται. Δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, ένα να προσθέσω μόνο. Η μελέτη για την ε, από κοινού οικειοποίηση. Είναι μελέτη της ομάδας εργασίας. Αλλά έτσι μπαίνουμε σε μια άλλη διάσταση που προτείνουμε εμείς την πρότασή μας. Ζητώ από τους συναδέρφους να υπερψηφίσουν. Πιστεύω ότι τα δύο που ζητάμε είναι συμπληρωματικά και αξίζουν τον κόπο να πρικοδοτηθούν με τόσα ζήτηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δίνουν προστιθέμενη αξία. ID δεν έχω κανέναν. Σωστά. Ωραία. Οπότε για το ECR ο κύριος Έπινγκ που δεν είναι εδώ. Κανείς εκ μέρους του. Οπότε φτάνω στον κύριο Γκούσμαν. Γκουε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο. Συγχαίρω τον εισηγητή που συμπεριέλαβε πολλές σημαντικές πτυχές. Θα δούμε τι θα γίνει με τις τροπολογίες για τα συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Η θέση μας είναι ότι τουλάχιστον δύο από τις συμβιβαστικές λύσεις υποστηρίζουν κάποιες θέσεις κάπως αντιφατικές, γιατί ο εισηγητής ήθελε να συμπεριλάβει τροπολογίες που είχαν διαφορετικούς στόχους. Η θέση μας θα καθοριστεί για το τι θα γίνει στην ψηφοφορία, ανάλογα με το τι θα γίνει και με τα αριθμητικά στοιχεία. Ευχαριστώ. Ζιγκφρίντ, έχει τον τελευταίο λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τους προς τον Σβέν Γκίγκολντ ε, για τον προϋπολογισμό για τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές. Καταρχήν, η αναθεώρηση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών δηλώνει ότι η ανάληψη των νέων αρμοδιοτήτων ε, ε, θα έχει χαμηλότερη απορρόφηση, γιατί πάντοτε είναι χαμηλότερη απορρόφηση από ό,τι φανταζόμαστε. Δεύτερον, ο συνολικός προϋπολογισμός μαζί με τις συνεισφορές του προϋπολογισμού είναι υψηλότερος από τον περσινό. Ε, δηλαδή τα υπόλοιπα έσοδά τους και η συνεισφορά του προϋπολογισμού ε, τελικά είναι υψηλότερο ποσοστό. Επειδή έχουν αυξηθεί ε, οι τα υπόλοιπα έσοδα θα είναι ο συνολικός του προϋπολογισμός υψηλότερος παρότι ο προϋπολογισμός της κοινότητας είναι στο ίδιο επίπεδο. Αυτά είναι τα δικά μου σχόλια. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και περιμένω την ψηφοφορία με μεγάλο ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε, Ζίγκφριτ. Ολοκληρώσαμε και αυτό το σημείο. Τώρα έχουμε και κλεισμένων των θυρών τη συνεδρία των συντονιστών. Μάρκους, θέλω να σε ρωτήσω. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο εναλλακτικέ λύσει. Μπορούμε να φύγουμε όλοι και να μείνουν οι συντονιστέ ή να πάνε οι συντονιστέ κάπου αλλού. Λοιπόν, ας φύγουμε όλοι οι υπόλοιποι και ας μείνουν οι συντονιστές στην αίθουσα και θα επανέλθουμε σε μισή ώρα για την ψηφοφορία. Θα γίνει τώρα η συνεδρία των συντονιστών.